ευχαριστώ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

Καλημέρα σας. Προτείνω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε ήδη ένα τέταρτο καθυστέρηση και γι' αυτό προτείνω να ξεκινήσουμε με την ημερήσια μας διάταξη. Έχουμε πολλά θέματα. Καλωσορίζω φυσικά όλους εσάς, όλους όσοι θα λάβουν το λόγο και θα σας παρουσιάσω τον κατάλογο των ομιλητών στη συνέχεια. Και θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για την απουσία του Αντιπροέδρου που αντικαθιστά εδώ ο κύριος Απτουλά Χασάν Κράισι, ο οποίος δεν εξασφάλισε την θεώρηση διαβατηρίου, τη βίζα εγκαίρως για να μπορέσει να έρθει στη σημερινή μας συνεδρίαση. Λυπούμε βαθύτατα γι' αυτό και το επεσήμανα ήδη στον πρεσβή Κυριέλα, ο οποίος όμως θα μας πει και δύο λόγια από ό,τι φαίνεται αργότερα. Ο Ρομπέρτ Ελπικά δεν ξέρω που είναι. Ριντμπερκ, δεν ξέρω που είναι, θα έρθει όμως. Για την ημέρη σε διάταξη παρακαλώ. Θέλετε να απαντήσετε μετά, να κάνετε την παρατηρήση σας μετά, για να μην χάσουμε χρόνο. Για να καταγραφείστε πρακτικά, βεβαίω. Βεβαίω και γι' αυτό με αυτό το θέμα ξεκινήσαμε. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, η έγκριση. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, έχετε παρατηρήσει. Είμαστε σύμφωνοι. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 15ης και 16ης Μαρτίου του 2009. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Καλώς. Σημείο 3. Αν μου επιτρέπετε, ανακοινώσει του Προέδρου. Της Προέδρου. Στη συνεδρίαση μας ε, και στην Ολομέλεια της 16ης Μαρτίου του 2009 ακούσαμε, από ό,τι θα θυμάστε, την Συμπρόεδρο της Ένωσης για την ε, Μεσόγειο σε μια έκτακτη συνεδρίαση. Είχαμε μάλιστα και τους Υπουργούς Αμπουγκάιτ και Μπερνάρ Κουσνέρ παρόντες με μια συνεδρίαση στην οποία έγινε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων εκφράστηκαν θέσεις και απόψεις. Έκτοτε λοιπόν έλαβε χώρα η συνάντηση του Προεδρείου στο Αμάν στις 4 Ιουλίου και το Προεδρείο υιοθέτησε μια διακήρυξη για το η Μέση Ανατολή. Διακήρυξη που θα δείτε στους φακέλους σας. Με την οποία διακήρυξη επαναβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του το Προεδρείο ότι θα συνεχίσει μέσω της κοινοβουλευτικής εργασίας της προσπάθειας για συμβολή στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώνει την πεποίθηση ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την ενεργό εμπλοκή όλων των παραγόντων της περιοχής, με την περάτωση των βιοπραξιών και πάνω απ' όλα με την ανάπτυξη μέτρων που θα εξασφαλίσουν εμπιστοσύνη στην ε, περιοχή και πάνω απ' όλα με πρώτη απόλυση ε, την πάυση της ε, πολιτικής των επικισμών της Ισραηλινής κυβέρνησης, την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνη και ειρήνης στην Δυτική Όχθη και τη Γάζα και την ανάπτυξη ενός μακροχρόνιου σχεδίου ειρήνης. Και θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα μέσα τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και τους Παλαιστινίους να συμβιώσουν στο μέλλον σε ειρήνη και ασφάλεια. Αυτές οι <clears throat> θεμητές επιθυμίες, αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζουμε να μπορέσουν να εγκριθούν σύντομα έτσι ώστε να καταγράψουμε ε, τις ε, θέσεις αυτές ως ε, συμπεράσματα σε μια διαδικασία ειρήνης για τη Μέση Ανατολή. Επίσης, η Πολιτική Επιτροπή θα πρέπει να συζητήσει, όπως είπαμε, θέματα που είχαν προβλεφθεί από το Μάρτιο του 2009 και εν ώψη τη ημερήσια διάταξη του Μαρτίου του 2010. Και έτσι σήμερα θα γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα δύο κύρια θέματα, δηλαδή τη διαδικασία τη Βαρκελόνη και την Ένωση για τη Μεσόγειο, θέμενη αξία που προσφέρει στην ανάπτυξη τη ε, περιοχή αυτή. Και δεύτερο θέμα, σεβασμό των θρησκευτικών ε, απόψεων και πεπιθήσεων θα γίνει άλλωστε σήμερα το απόγευμα η παρουσίαση των τοποθετήσεων από του ομιλητέ μα και θα ήθελα να του ευχαριστήσω γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι παρεμβάσει του. που θα συζητήσουμε το απόγευμα όπω είπα. Η προσεχή συνεδρία του Προεδρείου προβλέπεται για τι 20 Νοεμβρίου στο Κάιρο. Και φυσικά θα σα ενημερώσω ε, για τι οποίε αποφάσει ληφθούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, προ σήμερα μα είναι να κάνουμε μακροχρόνιο προγραμματισμό των εργασιών μα. Θα δείτε λοιπόν εδώ το χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων της Πολιτικής Επιτροπής για το 2010. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ε, Πολιτικής Επιτροπής ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ε, δείχνουν ότι δεν μπορούμε να ξεπερνούμε τις τέσσερις αναέτος συνεδριάσεις του 2010. Έχουμε λοιπόν τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο στο περιθώριο της Ολομέλειας, τον Ιούνιο και μετά το Σεπτέμβριο συνεδριάσεις. Και εν τέλει αγαπητοί συνάδελφοι υπενθυμίζω ότι από τη μία και μετά θα σας προσφέρουμε γεύμα στο ισόγειο του Κοινοβουλίου, στο σαλόνι των βουλευτών. Για δε τις τη διερμηνία έχουμε αγγλικά, γαλλικά, ε, ιταλικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, αραβικά, εβραϊκά και τουρκικά. Ε, και προτείνω να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Και θα συστήσουμε παρουσία του κυρίου Ρίτπερκ, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επικεφαλής του Τμήματος Μέση Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Σουηδικού Υπουργείου των Εξωτερικών, με την ευκαιρία της Σουηδικής Προεδρίας, του κυρίου Ραν Κουριέλ, πρέσβη του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της κυρίας Λίλα Σαΐντ, γενικής εκπροσώπου ε, απεσταλμένης της Παλαιστίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια θα ε, συζητήσουμε για τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρήνη, παρουσία της κυρίας ε, Mary T. Curtin, αναπληρώτριας Υπουργού των Πολιτικών Υποθέσεων και σύμβουλο στην, ε, στην Αμερικανική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθούμε και στα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η κατάσταση στην περιοχή είναι διαρκώς ε, λεπτή, ευάλωτη και ε, επικίνδυνοι και δεν έχουν καθόλου βοηθήσει τα τελευταία γεγονότα στην ε, διευκρίνηση των ε, καταστάσεων. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις σήμερα εδώ και παρά τις σαφείς δεσμεύσεις του Προέδρου Ομπάμα των ΗΠΑ η ειρηνευτική διαδικασία ακόμη βρίσκεται σε αδέξοδο και κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης των επικισμών. Πρόσφατη μελέτη του Transatlantic Trade του 2009 δείχνει ότι 77% των Ευρωπαίων πλέον υπεστήριξαν τον πρόεδρο Ομπάμα στις ε, διεθνείς του πρωτοβουλίες ενώ ήταν μόνο 18% εκείνοι οι οποίοι υπεστήριξαν την ε, ε, εξωτερική πολιτική του κυρίου Μπούς το 2008. Αναμένουμε λοιπόν τη κυρία Κέρτιν με αδημονία την παρουσίαση των πρωτοβουλειών των ΗΠΑ στην περιοχή και κυρίως ύστερα από την πρόσφατη επίσκεψη του George Mitchell, Αμερικανού απεσταλμένου στη Μέση Ανατολή. Όλοι μας παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον ε, την ε, περιοδία της κυρίας Χίλαρη Κλίντον ε, στην Μέση Ανατολή και το Μαρόκο πρόσφατα και τη συναντήσεις με τους υπουργούς των εξωτερικών από τα αραβικά κράτη. Πριν από δύο εβδομάδες οι Ισραηλινές πηγές μιλούσαν για μια άμεση επανάληψη των συνομιλιών, πράγμα το οποίο όμως αμφισβήτησε, διέψευσε καλύτερα ο Παλαιστίνιος αντιπρόσωπος το οποίο όμω καταδίκασε ταυτόχρονα και την αδιαλαξία των Ισραηλινών στην, ε, στην υπόθεση αυτή. Από τον Μαχμούτ Ταμπά, ακούμε ότι 24 Φεβρουαρίου αναμένονται εκλογέ στην ε, Παλαιστίνη και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική πρωτοβουλία θα πρέπει αποκλειστικά να συνδεθεί με την περάτωση των, ε, με την διακοπή των επικισμών. Και προβλέπεται, από ό,τι φαίνεται, μια πρόθεση για ανακήρυξη Παλαιστινιακού κράτους σε δύο χρόνια. Βλέπετε λοιπόν στη φακέλους σας ε, την βούληση για προστασία των ε, πιο αδύναμων για την ανάπτυξη μιας ειρήνης ε, διαρκούς και πολιτικής ανεξαρτησίας και μόνο η συμφιλίωση μεταξύ ΧΑΤΑ και ΦΑΤ. Φατάχ, ε, Χαμάς και Φατάχ σε επίπεδο Παλαιστινιών θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ενότητα των Παλαιστινιών. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνουμε τις ενδοπαλαιστινιακές συνομιλίες με τις τρεις βασικές αρχές που που έχει υιοθετήσει η τριμερής, δηλαδή αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, αποδοχή των προηγούμενων συμφωνιών και αποκήρυξη της βίας. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις οποίες δεσμεύεται να λάβει η Χαμάς ως προς το σεβασμό αυτών των ε, όρων. Πλην όμως δεν θα πρέπει και να λησμονούμε την ανθρωπιστική κατάσταση, την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στην ε, ε, λωρίδα της Γάζας, την ανάγκη να ανοιχθούν δύο διπεράσματος που θα διευκολύνουν την ανοικοδόμηση κατεπηγόντως, πράγμα το οποίο άλλωστε έχει επιβεβαιώσει και ο κύριος Άντερς Λίντεν, Σουηδό πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη 14 Οκτωβρίου. Η διαρκής λοιπόν ε, επικοινωνία με τη Λωρίδα τη Γάστα θα πρέπει να εξασφαλιστεί χάρη ε, στο ψήσιμο 1860 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για άμεσο άνοιγμα και ανεφόρον άνοιγμα των διόδων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μετάβαση τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λόρδια της Γάζας. Άλλοι λόγοι κρίσεως επίσης, η συνέχεια που θα πρέπει να αποδοθεί στην έκθεση Goldstone, δηλαδή τη μελέτη για τους λόγους αυτής της κρίσης στη Γάζα που ε, ανέπτυξα ε, με πρωτοβουλία της Υποεπιτροπή των ε, Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των ΕΕ. Εθνών. Θα δείτε στα έγγραφά σα τα συμπεράσματα αυτή τη έκθεση, καθώ και έγγραφο του Υπουργείου των Εξωτερικών του Ισραήλ με τίτλο αρχική ανταπόκριση στην ερευνητική αποστολή στη Λόρδα της Γάζας. Η Γενική Συνέλευση των Εθνών πρόκειται να συζητήσει την έκθεση αυτή το Νοέμβριο εφέτος και εμείς αγαπητοί συνάδελφοι κατά την ανταλλαγή απόψεων θα θίξουμε και το θέμα αυτό. Και τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κύριε Ρίτπερκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω που οργανώσατε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για ένα θέμα το οποίο είναι προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής αυτής της Προεδρίας και θα παραμείνει τέτοιο και μετά το πέρας της Προεδρίας μας. Θα μιλήσω για τις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Προεδρίας και θα σας πω ποια είναι η εκτίμησή μας για την κατάσταση της ειρηνευτικής διαδικασίας της Μέσης Ανατολής. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από διάφορες αντιθέσεις και αντιφάσεις. Έχουμε μία έντονη εμπλοκή των Αμερικανών και όμως η διαδικασία ε, έχει βουλιάξει και δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Ε, η αντιμετώπιση του ενός ε, από τον άλλο χαρακτηρίζεται από δυσπιστία. Υπάρχει επίσης αυξανόμενη διεθνής επίκριση. Από την ε, πλευρά των Παλαιστινίων υπάρχουν έντονες, ε, έντονοι διχασμοί και υπάρχουν σοβαρές ε, δυσκολίες. Υπάρχει μια σχετική απουσία ε, διευρυμένης βίας και όμως οι εντάσεις είναι πολύ έντονες, προφανώς στην Ιερουσαλήμ, αλλά κατά καιρού και στη Λωρίδα της Βάζας, στα σύνορα με το Λίβανο και αλλού όμως. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία ε, εμπεριέχει τα ψήγματα των, ε, της αλλαγής αλλά και τους κινδύνους. Οι προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η πανέναξη των διαπραγματεύσεων, η ενδυνάμωση του Προέδρου Αμπάς και η εστίαση της όποιας κατάστασης επιτόπους και στη λόγια της, Γάζας. Ο συντονισμός με τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικός και ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για αυτόν τον σκοπό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει ε, υποστήριξη για την, ε, τις προσπάθειες των ΗΠΑ για να υπάρξει μια δικρατική λύση. Ε, είπαμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος το οποίο θα ζει δίπλα-δίπλα με ασφάλεια και ειρήνη με το κράτος του Ισραήλ θα θέλαμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ε, με ένα σαφή στόχο και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Ε, η Αμερικανική ηγεσία θα πρέπει να υποστηρίξει και το κουαρτέτο και την αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις και πολιτικά αλλά και με συγκεκριμένες δράσεις. Η προσπάθεια συνεχίζεται, ιδίω το τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε την οικοδόμηση ενό Παλαιστινιακού κράτου και να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε για να υπάρξει μια πλήρη επίλυση τη Άραβο-Ισραηλινή διένεξη. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία ε, τη οικοδόμηση ενό Παλαιστινιακού κράτου. Είναι μια διαδικασία παράλληλη με τι διαπραγματεύσει, αλλά και είναι ένα επικοδομητικό τρόπο ε, για να υπάρξει μια πολιτική λύση αν υπάρξει πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Εμείς στην ομάδα των δωρητών έχουμε πάρει μια ηγετική θέση. Ε, θέλουμε να προωθήσουμε, την, να, να σταματήσει η κατοχή και να συνεχίσουμε την παροχή βοήθειας Μετά την Υπουργική Τρόικα και τον πολιτικό διάλογο, τώρα εξετάζουμε το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε επίσημες σχέσεις με την Παλαιστίνη. Καλωσορίζουμε το αίτημα του Πρόεδρου Αμπάς για εκλογές στην Παλαιστίνη, στην δυστική Ιερουσαλήμ, στη Γάζα και ενθαρρύνουμε την Παλαιστινιακή συμφιλίωση πίσω από τον Πρόεδρο Χαμπάς και Υποστηρίζουμε την Αίγυπτο και τις διαμεσολαβητικές της προσπάθειες. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεραστούν οι εσωτερικές διαμάχες ε, αν θέλουμε να υπάρξει ενότητα και ένα, στα πλαίσια ενός Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις εκλογές και για την ε, ανοικοδόμηση της Γάζας. Επίσης είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εξουσία της Χαμάς στην Γάζα ε, συνοδεύεται από πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δράσεις ε, με σκοπό να ε, μην υπάρξει καμία πολιτική εναλλακτική λύση. Επίσης θα εκφράσουμε στο διάλογό μας με την Παλαιστινιακή Αρχή όλες τις ανησυχίες που έχουμε για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι σχέσεις μας με την Παλαιστινιακή Αρχή είναι καλές ε, τον Ιούνιο συναντήθηκε το Συμβούλιο Σύνδεσης και έχουμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με βάση το σημερινό σχέδιο δράσης, που είναι ίσως ε, το πιο προχωρημένο που είχαμε ε, με οποιοδήποτε νότιο γείτονα. Γι' αυτό στις Βρυξέλλες θα υπογράψουμε μια νέα γεωργική συμφωνία. Θα υπογράψουμε προσεχώς επίσης μια συμφωνία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων. Στο πολιτικό τομέα υπάρχουν έντονες διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα και σε αυτή την Προεδρία ήδη είχαμε επαφές σε επίπεδο ομάδων εργασίας και ελπίζουμε να υπάρχει πλήρης πολιτικός διάλογος. Αγαπητή Πρόεδρε, η διεθνής υποστήριξη, η προσπάθειά μας και τα θετικά βήματα από πλευράς Ισραήλ έχουν βοηθήσει στο να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στη Δυτική Όχθη. Ε, και υπάρχουν και ορισμένες οικονομικές επιπτώσεις ε, επιτόπου. Θα πρέπει να προχωρήσει η δουλειά όμως ακριβώς για αυτό το σκοπό του κουαρτέτου και άλλων. Αυτές οι βελτιώσεις δεν αρκούν όμως. Είναι ασθενής η θέση της Παλαιστινικής Αρχής, επεκτείνονται οι επικισμοί και υπάρχει όλο και μεγαλύτερος διαχωρισμός των βασικών εταίρων στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τις ανησυχίες της κατ' επανάληψη για τις εξελίξεις επιτόπου, ιδίως την συνεχιζόμενη απομόνωση της Γάζας, της τις προκλήσεις στην Ιερουσαλήμ και την εξάπλωση των επικισμών. Η, η Γάζα είναι μια καταστροφή που περιμένει να ολοκληρωθεί. Αυτή η πολιτική απομόνωση έχει σοβαρότατες ανθρωπιστικές συνέπειες και ενώ ε, κερδίζουν από αυτή την ιστορία ε, οι υπεύθυνοι των τούνελ, στην πραγματικότητα οικονομικά αποδυναμώνονται οι κάτοικοι της Γάζας. Θα πρέπει να ανοίξει τα περάσματα της Γάζας. Ε, έχουμε θέσει αυτό το θέμα σε πάρα πολλές επιστολές ε, προς την κυβέρνηση του Ισραήλ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οι Ισραηλινοί δεν ανταποκρίνονται και αυτό είναι απαράδεκτο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλα διαβήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Προ την κυβέρνηση του Ισραήλ και προς την Παλαιστινιακή Αρχή έχουμε εκφράσει τι ανησυχίε μας για την ασταθή κατάσταση στην Ιερουσαλήμ και για τις προκλήσεις που υπάρχουν. Η Ιερουσαλήμ είναι ένα τεράστιο θέμα ε, για να υπάρξει επίλυση. Δεν υπάρχει περίπτωση ε, δημιουργία της λύση λύσης ε, χωρίς να επιληθεί το θέμα της Ιερουσαλήμ. Επίσης, οι εξώσει, ε, η επέκταση των επικισμών, όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να αποφευθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έκκληση στο Ισραήλ να σταματήσει τις ε, δραστηριότητες σε επίπεδο ε, επικισμών και να διαλύσει όλα τα προκεχωρημένα φυλάκια που ύψωσε μετά το Μάρτιο του 2001. Αγαπητοί φίλοι, η διαδικασία στη Μέση Ανατολή βασίζεται ε, στο διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η θέση που λάβαμε και πρόσφατα σε διάφορες συζητήσεις που κάναμε στη Νέα Υόρκη και στη Γενέβη με βάση την έκθεση Goldstone και, το... και συζητήσεις για το τείχος ε, της Λοδιάς της Γάζας. Έχουμε θεσμευτεί να λάβουμε υπόψη σοβαρά αυτή την ε, έκθεση. Η προτεραιότητά μας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μη συνεχιστεί αυτή η ατιμορρησία. Επομένως θα θέλαμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να ξεκινήσουν ανεξάρτητες και αξιόπιστες έρευνες σε οποιασδήποτε παραβιάσεις ε, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τα διεθνή πρότυπα. Καταληκτικά, Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία μια περιφερειακή προσέγγιση στην σύγκρουση ε, Ισραήλ και Αράβων. Για να υπάρξει βιώσιμη λύση, θα πρέπει να υπάρξει παράλληλη πρόοδο ε, σε επίπεδο σχέσεων Ισραήλ-Λιβάνου ε, και Ισραήλ-Συρίας. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε ένα σημαντικό βήμα γιατί ε, με τη Συρία προχωράμε σε μια συμφωνία σύνδεσης. Έχουμε στενές επαφές με το Λίβανο και υποστηρίζουμε την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1701 ως στρατηγικό μέσο για την ε, περιφερειακή ασφάλεια. Επιπλέον, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ε, αποφασιστική στο διμερή διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μέρη της ε, περιοχής και σε επαφές που έχουμε με, την, με τον Αραβικό Σύνδεσμο, με οργανώσεις των Αραβικών χωρών και στο εσωτερικό βέβαια της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρίτμπεργκ. Τώρα ο πρέσβης Κυριέλ θα έχει το λόγο. Θέλω μόνο να σας πω ότι τα μέλη της Κνεσέτ δεν είναι παρόντα γιατί δεν έχουν ακόμα οριστεί. Αυτό μου είπε ο κύριος πρέσβης. Λοιπόν, κύριε πρέσβη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαϊφή. Θέλω να καλωσορίσω εδώ και τον κύριο Μπέλα Μπέλα που ήταν ε, πριν ε, συναδερφός μου. Του συναδέρφους επίσης ε, Ρίτμπεργκ, Ραΐ και το υπόλοιπο Προεδρείο εδώ. Ειλικρινά για μένα είναι μεγάλη χαρά που μπορώ και βρίσκομαι εδώ μαζί σας και που μπορούμε να έχουμε καρποφόρες συζητήσεις εδώ σήμερα το πρωί. Υποστηρίζω το στόχο όλων, δηλαδή να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Καταλαβαίνω ότι και εβραϊκά υπάρχει μετάφραση και από εβραϊκά, οπότε θα μου επιτρέψετε να περάσω στη μητρική μου γλώσσα. Ελπίζω οι συζητήσεις μας να μπορέσουν να είναι καρποφόρες. Πιστεύω ότι για όλους εσάς που παρακολουθείτε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ξέρετε ότι ο πρώτος, ο κύριος στόχος είναι στόχος όλων όσοι θέλουν να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με μας και ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή είναι προ το συμφέρον όλων, και του Ισραήλ και της Αμερικής και της Ευρώπης, όπως εξάλλου το ακούσαμε πριν από λίγο. Συνεπώ είναι προ το συμφέρον και των Παλαιστινίων. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στην ειρήνη χωρίς διαπραγματεύσεις για την ειρήνη προηγουμένω και όπως ξέρετε προσπάθειες κάνουμε, προσπάθειε σοβαρέ. Η Αμερικανική κυβέρνηση για παράδειγμα η Υπουργό Εξωτερικών Κλίντον που ήταν στο Ισραήλ ε, πριν από λίγο, ο Μίτσελ επίσης, ο Νιωτανάου το είπε και θα πάει στην Ουάσιγκτον και ο Υπουργό Άμυνα, η Κλίντον μετά πήγε στο Μαρόκο. Νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει. Είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ θέλει να ξαναρχίσουν σήμερα, τώρα, αμέσω, χτε, αν είναι δυνατόν, οι διαπραγματεύσει. Τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα για όλους όσοι βρίσκονται εδώ σήμερα και χωρίς προϋποθέσεις. Όλα τα θέματα μπορούν να συζητηθούν γύρω από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτός είναι και ο κύριος στόχος μας. Αν να δούμε τα πράγματα ιστορικά κάπως, ξέρουμε ότι έχουμε εδώ και Αιγυπτίους και Ιορδανούς και ξέρουμε ότι εδώ και 30 χρόνια το Ισραήλ έχει φύγει από το ΣΥΝΑ, έχει επιστρέψει εδάφη στην Ιορδανική κυβέρνηση και όλα αυτά προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη με τους γειτονές μας. Αυτό είναι βασικό και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο και με τους Παλαιστίνιους γειτονές μας. Εξάλλου, φύγαμε από τη λωρίδα της Γάζας το 2005. Το Ισραήλ άδειασε εντελώς τη λωρίδα της Γάζας και από στρατιώτες αλλά και από πολίτες διότι ε, τα σπίτια εκεί τα διάσαμε. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια θετική διαδικασία στην Γάζα. Δεν υπάρχουν Ισραηλινοί πια στη Γάζα. Δυστυχώ, βέβαια αυτά που έγιναν στη Γάζα μετά ε, δεν αποτελούν για ένα θετικό παράδειγμα για το πώς πρέπει να έχει κατάσταση επιτόπου, ούτε είναι κάτι θετικό για την κοινή γνώμη στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργό Νιωταχάου και το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις που να περιλαμβάνουν όλα τα θέματα βάσει της λύσης δύο κράτη για δύο λαούς. Διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στο τέλος της σύγκρουσης και που θα οδηγήσει στο τέλος των, ε, της κατοχής. Νομίζω λοιπόν ότι με το πολιτικό χρώμα της ελληνικής κυβέρνησης και αν δούμε την κοινή γνώμη στο Ισραήλ, τον κόσμο, την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου στο Ισραήλ, ε, λοιπόν όλοι αυτοί θέλουν να υπάρξει πολιτικά χωρισμός με τους πολυστηνίους. Θέλουν να φτάσουν στη λύση δύο κράτη για δύο λαούς. Και πιστεύω ότι εφόσον οι Ισραηλινοί έχουν κάποια αμφιβολία ή έχουν αμφιβολίες, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Τότε οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να οδηγήσουν στην διατήρηση του χαρακτήρα του Ισραήλ ως ένα εθνικό Ισραηλινό κράτος και δεύτερον να μην αφισβητηθεί η ασφάλεια του Ισραήλ. Είναι λοιπόν αναγκαίο να έχουμε κάποιες διαβεβαιώσεις για αυτό το θέμα. Να διατηρηθεί λοιπόν ο χαρακτήρας, ο Ισραηλινός χαρακτήρας του Ισραήλ και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους. Να μην πάμε πίσω όπως έγινε με το πείραμα της Γάζας που ήταν τόσο ατυχές. Μάλιστα, αν θυμόσαστε την απόφαση του 47 του Ισραήλ για την κατανομή ε, της γης του Ισραήλ σε δύο κράτη, θέλαμε ένα εβραϊκό κράτος και ένα αραβικό κράτος. Από το 47, έτσι. Δεν πρόκειται για ένα Ισραηλινό και μουσουλμανικό κράτος. Το ευρωαϊκό κράτος λοιπόν ήθελε τον εθνικό χαρακτήρα και όχι τον θρησκευτικό χαρακτήρα του κράτους και αυτό ακριβώ ζητάει το Ισραήλ και σήμερα. Και νομίζω λοιπόν ότι κάθε λογικός άνθρωπος ξέρει ότι όταν μιλάμε για δύο κράτη μιλάμε και για μια συγκεκριμένη ερμηνεία, δηλαδή δύο κράτη για δύο λαούς που και για τους Ισραηλινούς αλλά και για όλους νομίζω σημαίνει ένα Παλαιστινιακό κράτος το οποίο θα εκφράζει την αυτοδιάθεση, την εθνική αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων και το Ισραήλ την αυτοδιάθεση του λαού του Ισραήλ στη γη του. Αυτό σημαίνει δύο κράτη για δύο λαούς. Μέχρι σήμερα δεν έχω την αίσθηση ότι έχουμε πάρει σαφή και ξεκάθαρη απάντηση σε αυτήν τη θέση του Ισραήλ. Όταν λοιπόν λέμε δύο κράτη πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε. Γιατί η ερμηνεία του Ισραήλ που εμένα μου φαίνεται απόλυτα θεμητή είναι αυτή η συγκεκριμένη που σημαίνει κάποια πράγματα βέβαια για το δημογραφικό, για παράδειγμα σκέλος. Οι λίγοι ε, Άραβες που θα ζουν στο Ισραήλ, όπως και μέχρι σήμερα, θα έχουν όλα τα δικαιώματα, όπως οποιοδήποτε δημοκρατικό κράτος. Αλλά η έκφραση πάντως εθνική ταυτότητα πρέπει να έχει να κάνει με το Παλαιστινιακό κράτος. Νομίζω λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν σημαντικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα σύνορα, οι επικοικισμοί, ε, το εδαφικό, το αεροσόλυμα, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Πάντως εδώ σήμερα, σε αυτή την αίθουσα, οφείλω να σας πω ότι πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα απ' όλα μια ατμόσφαιρα ειρήνης. Μια ατμόσφαιρα η οποία θα επιτρέψει να διασφαλίσουμε για την κοινή γνώμη τόσο του Ζήλου όσο και της Παλαιστίνης ότι πραγματικά υπάρχει πρόθεση να φτάσουμε στην ειρήνη. Δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν είναι αυτό το αίσθημα που εισπράττει ο Ζελινός λαός. Δεν υπάρχει πάντα. Ακόμα και εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο, δεν υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα ειρήνης. Μερικές φορές φεύγω από εδώ και τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι ναι, δεν υπάρχει θέληση από την άλλη μεριά πραγματικά να φτάσουμε στην ειρήνη, αλλά υπάρχει διάθεση να κατηγορήσουν το Ισραήλ, να τα βάλουν με το Ισραήλ, να καταγγείλουν το Ισραήλ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρξει και εδώ αυτό ο θετικό τόνο, αυτή η θετική ατμόσφαιρα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί είναι κάτι που αποτελεί πλήρω μέρο μια ειρηνευτική διαδικασία. Το πρόβλημα ανάμεσα στο Ισραήλ και του Παλαιστινίου δεν είναι το μόνο πρόβλημα, η σύγκρουση αυτή δεν είναι η μόνη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξάλλου. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχουν οι ακραίοι και οι μετριοπαθείς στη Μέση Ανατολή και αυτή είναι η σύγκρουση. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που θέλει την ειρήνη πρέπει να στηρίξει τους μετριοπαθείς στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να απομονώσουμε τους ακραίους που εμποδίζουν κάθε δυνατότητα πρόσβαση στην ειρήνη. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες να αναφερθώ στο Ιράν. Το Ιράν φυσικά είναι κεντρικό ζήτημα στη Μέση Ανατολή και τα πράγματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, είτε το θέλουμε είτε όχι. Η δυνατότητα να φτάσουμε στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αλλά το Ιράν παρεμβαίνει εκεί που θέλει πυρηνικά. Κύριε Πρέσβη Ρίτμπερ, συμφωνώ μαζί σας με αυτά που είπατε για το ότι δηλαδή οι καλές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρώπη υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε υπογράψει μεταξύ μας από το 1975 Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Ο Εβραϊκός λαός και η Ευρώπη έχουν δεσμούς εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν βέβαια και σκοτεινά σημεία, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ θετικά σημεία στην ιστορία των μεταξύ μας ανεξάρτητα με το τι συμφωνίες ε, υπάρχουν ή θα υπάρχουν ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρώπη, οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν ένα διάλογο σε επίπεδο ενηλίκων, υπεύθυνο, και ακόμα και αν δεν συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, γίνεται αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να κόβουμε όλες τις γέφυρες, δεν πρέπει να κόβουμε τις επαφές κάθε φορά που υπάρχει διαφωνία για το ένα ή το άλλο θέμα. Ένα μέρος των συμφωνιών στις οποίες αναφερθήκατε, γεωργικές για παράδειγμα, είναι διμερείς συμφωνίες. Χρησιμεύουν και για την Ευρώπη και για το Ισραήλ. Είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Οπότε η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ είναι κάτι πάρα πολύ θετικό από πλευράς του Ισραήλ. Εξάλλου το Ισραήλ έχει αλλάξει τη θέση του απέναντι στην Ευρώπη. Τα τελευταία, τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε ότι θέλουμε όλο και πιο στενές σχέσεις με την Ευρώπη, Ευρώπη που στηρίζει τη διαδικασία ειρήνευσης. Όλες οι πλευρές στην περιοχή χρειάζονται τη στήριξη ολονών σε ολόκληρο τον κόσμο για να λυθεί η σύγκρουση αυτή, τόσο από πλευρά της Αμερικής όσο και από πλευρά της Ευρώπης. Η Ευρώπη μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Θα αναφερθώ σε άλλα θέματα αργότερα στη συζήτηση, αλλά για να απαντήσω σε αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, Θέλω να μιλήσω σε κάτι στο οποίο αναφερθήκατε, Πρόεδρε Σέφη, για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Οι δύο προς τη Γάζα είναι ανοιχτές για ανθρωπιστική βοήθεια. Ακόμα και κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τη αρχή της χρονιάς, οι δύο αυτοί ήταν πάντα ανοιχτες Και αυτή είναι η διαφορά. Άλλο οι δύο ανθρωπιστικης βοηθειας και άλλο οι οικονομικες σχεσεις οι κανονικες ανάμεσα στην ε, Γκάζα και το Ισραήλ. Αυτές οι δύο δι, είτε πρόκειται για πρόσβαση ανθρωπιστικού υλικού, τρόφιμα, καυσίμων κτλ, παραμένουν ανοιχτές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άλλη ανθρωπιστική συζήτηση λοιπόν και άλλο οικονομικές σχέσεις, ισορροπημένες κανονικές σχέσεις ανάμεσα σε μία ε, μονάδα που είναι τρομοκρατική και ζητά την καταστροφή του Ισραήλ και άλλο ε, το κράτος που βρίσκεται από την άλλη πλευρά. Τώρα για τους επικισμούς μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο και σίγουρα θα τεθεί και κατά τη συζήτηση, αλλά δεν θα είναι το μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Το Ισραήλ το έχει δείξει και από το παρελθόν ότι οι επικισμοί δεν είναι το εμπόδιο στην ειρήνη. Έχουμε ε, στο Σινά, για παράδειγμα, καταστρέψει του επικισμού εκεί για να έχουμε συμφωνία με την Αίγυπτο. Έχουμε καταστρέψει επικισμού επίση στη Γάζα. Υπάρχουν τρομακτικές αλλαγές όσον αφορά τους ε, επικισμούς τον τελευταίο καιρό. Ο Νιατανάου τι είπε δίπλα στην Κλίτον του Δευτέρα ήταν ή την Τρίτη. Το είπα αυτό. Μπορούμε μερικές φορές να πάρουμε ένα θέμα και να το κάνουμε το κέντρο, τον πυρήνα της συζήτησης. Αλλά δεν είναι αυτό το κεντρικό σημείο στη συζήτηση. Δεν θα έπρεπε. Θα σας διαβάσω λοιπόν πραγματικά ο Νιτανιάου αυτή τη βδομάδα δίπλα στην ε, Υπουργό Εξωτερικών Κλίντον, στα αγγλικά δεν θα κτίσουμε νέους επικισμούς, δεν θα απαλωτριώσουμε γη για τους επικισμούς που φτιάχνονται τώρα. Είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε επικισμούς και τους ήδη υπάρχοντες, αλλά υπό τον όρο να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν κανονικά τις ζωές τους. Το θέμα των επικισμών και το θέμα των εδαφών και των συνόρων είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις και πρέπει να λυθούν με ειρηνευτική, προκειμένου να πετύχουμε την ειρηνευτική συμφωνία. Μπορούν να λυθούν αυτά τα θέματα πριν από τις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί να μπει αυτό σαν προϋπόθεση. Αυτά είπε ο Νιατανάου. Αυτή ήταν η απάντησή του. Τώρα για τη μελλοντική συμφωνία, κυρίες και κύριοι. Εγώ πιστεύω και αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση, αν μου επιτρέπετε να έχω μία ως πρέσβης, ότι αν θέλουμε δύο κράτη, και πιστεύω ότι θα έχουμε δύο κράτη, το Παλαιστινιακό δίπλα στο Ισραήλ, δεν θα υπάρχουν επικισμοί στο Παλαιστινιακό κράτος. Και κατά πάσα πιθανότητα, παραπάνω από κατά πάσα πιθανότητα, το Ισραήλ θα μείνει με 20% του πληθυσμού του να είναι Άραβες Παλαιστίνοι. Αυτό θα γίνει όταν μιλάμε για επικισμούς. Λοιπόν, εγώ σαν μήνυμα λέω, ας καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ας ξεκινήσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος να καταφέρουμε να πετύχουμε την ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο τώρα παρακαλώ να λάβει η κυρία Γενική ε, κατασταλμένη της Παλαιστίνης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την Πολιτική Επιτροπή της Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης που μας επιτρέπει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της συσμευτικής διαδικασίας να λάβουμε το λόγο σε μια ανταλλαγή απόψεων. Και τώρα θα μιλήσω αγγλικά. Ίσως είναι πιο εύκολο για όλους. Ξεκινώντας, θα ήθελα προς τον Ισραηλό, συνάδελφο που ε, εκφράζεται την του για το ότι δεν είναι κατάλληλη η ατμόσφαιρα ή το κλίμα για την ειρηνευτική διαδικασία. Να πω ότι η παρουσία εδώ και του Δ. Αμπτάλα Αμπτάλ, επικεφαλή πολιτική επιτροπή, αλλά και τη ε, πρέσβεω, είναι μια πολύ ασυνήθιστη παρουσία για ε, ένα λαό που αγωνίζεται για την ελευθερία. Είναι πολύ σπάνια αυτή η ευκαιρία και την οφείλουμε στους Ευρωπαίους φίλους μας που μας επιτρέπουν να καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων καλύτερα σε, μια, σε ένα χώρο στον οποίο εκπροσωπούνται τόσο ευρωπαϊκές όσο και αραβικές χώρες. Ευχαριστώ ιδιαίτερως λοιπόν τους Ευρωπαίους οικοδεσπότες μας, την Πολιτική Επιτροπή της Ευρωμεσογειακής κοινοβουλευτική Διασπέσεως σκέψεως που μας δίνουν την ευκαιρία αυτή, διότι πλέον δεν βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ισραηλινούς για την ειρήνη. Σα υπενθυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσονται ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει. Οι διαπραγματεύσει μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη έχουν ξεκινήσει εδώ και 18 χρόνια και περισσότερο στη Μαδρίτη. Σας το υπενθυμίζω, διότι σε μερικές ημέρες θα χαιρετήσουμε την επέτειο της πτώσης του τείχου του Βερολίνου. Σα πενθυμίσω λοιπόν ήταν οι πρώτε διαπραγματεύσει που αναπτύχθηκαν μετά την κατάρρευση του τείχου, μετά δηλαδή την κατάρρευση του διχασμού τη διχοτόμησης Ανατολικό και Δυτικό Μπλοκ. όπω είπε και ο πρέσβη Ρούτσμπερκ, η προτεραιότητα για ειρήνη και ειρηνευτικές διαδικασίες ανά τον κόσμο δίδεται ιδιαίτερα στην Μέση Ανατολή που βρίσκεται άλλωστε και στο επίκεντρο στην καρδιά της ε, Μεσογείου. Οι διαπραγματεύσει ήταν και διμερεί αλλά και πολυμερεί ταυτόχρονα. Και θα ήθελα να πω ότι οι Παλαιστινοί δεν δίστασαν ποτέ να αναλάβουν την ευθύνη της άμεσης διαπραγμάτευσης παρά το γεγονός ότι δεν έχει περατωθεί η κατοχή τόσο στο Όσλο όσο και στην Ανάπολη συμμετέχαμε στις διαπραγματεύσεις χωρίς όμως να σημειωθεί πρόοδος των αντίον θα έλεγα ότι έχει μάλλον σημειωθεί οπισθοδρόμηση αν δούμε το τείχος το οποίο χτίζουν μέσα σε παλαιστινιακά εδάφη και όχι στα σύνορα οι Εβραίοι, εάν δούμε την επέκταση των επικισμών και αν δούμε την προσάρτηση της Ιερουσαλήμ. Πριν όμως εξακολουθούμε τις προσπάθειές μας γιατί θεωρούμε ότι είναι αυτός ο τρόπος ο καλύτερος για να δείξουμε στον κόσμο πόσο στρατευμένοι είμαστε στον αγώνα για την ε, ειρήνη. Στράτευση, κινητοποίηση, ταυτόχρονα εκφράστηκε και από τις πολυμερείς δομές, Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ τις προσπάθειές μας στη Μαδρίτη, τις προσπάθειές μας ιδιαίτερα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με όλα τα μέρη της, της τετραμερούς και ξεκινήσαμε, θα σημειώσω, με μια σειρά προσπαθειών, συμφωνιών, την οποία μόνο θα απαριθμίσω, γιατί θα πρέπει να θυμούμαστε ότι δεν μπορούμε με κάθε νέα Ισραηλινή κυβέρνηση να ξεκινάμε με ε, βάση μηδενική. Έχουμε ήδη την έβδομη κυβέρνηση από το Ισραήλ από τη στιγμή των τη εκείνη των διαπραγματεύσεων. Αν λοιπόν θέλετε κάθε φορά να ξεκινάμε σε μηδενική βάση, δεν θα φτάσουμε πουθενά ούτε στην ισραηλινο ειρήνη, ούτε και στην περιφερειακή ειρήνη. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων που συμφωνήσαμε διμερώς ήταν οι αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης. Στο Όσλο 2 το πέρας της κατοχής καταρχήν, τον, ε, το φιλοπορία, το νοδικό χάρτη όπως λέγεται, που ήταν μια πολύ καλή ε, προσέγγιση για παράλληλε δεσμεύσει, η υπενθύμηση των παραλληλών δεσμεύσεων και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω στον Πρεσβευτή Κυριέλ ότι υπάρχει δέσμευση για απόλυτο πάγωμα των επικισμών από πλευρά του Ισραήλ, ταυτόχρονα από την Παλαιστινιακή Αρχή δέσμευση για την καταπολέμηση τη ε, τρομοκρατίας. Όμω, θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχουν άλλε δύο πολύ σημαντικέ ε, δεσμεύσει μία την οποία ε, ε, ανέλαβαν τα αραβικά κράτη της αραβικής, του Αραβικού Συνδέσμου του 2002 και που επανέλαβε η Ισλαμική Οργάνωση 50 ε, και χώρες την ειρήνη μεταξύ των Αράβων με το Ισραήλ αλλά και τη δέσμευση της Ετραμερούς για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων του φύλου πορεία. Όλε αυτέ λοιπόν οι κινήσει ακολουθούν ουσιαστικά τι διαπραγματεύσει μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων αλλά δυστυχώ, από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε μόνοι μα να τα καταφέρουμε όλα αυτά και γι' αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι καθήκον μα είναι ω Παλαιστινιακή Αρχή, ω ηγέτε δηλαδή, του λαού μα, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και υπεύθυνα να στρεφόμαστε και να, απευθυνόμαστε προς την κοινή μας γνώμη. Δεν έχει μόνο το Ισραήλ κοινή γνώμη κυρία Πρεσβευτά αλλά και η Παλαιστίνη και ολόκληρος ο κόσμος και γι' αυτό η κοινή μας γνώμη μας ζητά να ε, απαντήσουμε πως είναι δυνατόν ένα χρόνο μετά την Ανάπολη η μόνη απάντηση του Ισραήλ να είναι μια επίθεση κατά μέτωπο κατά της λωρίδας του Ισραήλ που αποτελεί κομμάτι των κατεχωμένων Παλαιστινιακών εδαφών με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και υπενθυμίζω άμαχους κατοίκους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρομοκρατική δραστηριότητα όχι μόνο στη Γάζα αλλά και σε κάθε κατεχόμενο έδαφος γιατί, σε, γιατί η κατοχή εκτρέφει την τρομοκρατία. Δεν είναι όμως κομμάτι του Ισραήλ η Γάζα. Η Λόρδα της Γάζας είναι κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος το οποίο ζουν στο οποίο έλαβαν χώρα όχι μόνο οι πιο σοβαρές τραγικές και εγκληματικές δραστηριότητες επίθεσης ένα χρόνο μετά την ανάπολη πέρυσι αλλά και ταυτόχρονα ε, μπορεί εσείς να λέτε ότι υπάρχει πρόσβαση ανθρωπιστική στη γάζα αυτό ισχυρίζεστε εσείς αλλά θα σας πενθυμίσω ότι η ευρωπαϊκή ένωση πολύ καλό σας εταίρος κατά τα άλλα έχει δημοσιεύσει έχει καταγγείλει δημόσια το γεγονό ότι δεν μπορεί ούτε καν, όχι η ανθρωπιστική, ούτε καν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να περάσει στη Λόριδα τη Γάζα, αυτόν τον αποκλεισμένο πληθυσμό. Ε, υπάρχει επίση Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, νέα, νέο συσταθή επιτροπή, η οποία έχει μελετήσει την κατάσταση και η οποία απερίφραστα έχει καταδικάσει τι ε, εγκληματικέ σα δραστηριότητε, τι εγκληματικέ δραστηριότητε του Ισραήλ στη Λωρίδα τη Γάζα. Πρόκειται για την Επιτροπή Goldstone και θα ήθελα να ακούσω τι απαντήσει εκεί, γιατί είναι ευθύνη όχι μόνο κυβέρνηση του Ισραήλ, αλλά είναι ευθύνη σα και ω μέλους της κοινότητας των Ηνωμένων Εθνών, της διεθνούς κοινότητας. Πρέπει λοιπόν και ελπίζω η προσεχής ε, Γενική Συνέλευση να δώσει την ευκαιρία στο κάθε κράτος μέλος να εκφράσει τις θέσεις του και τις γνώμες του για αυτό το οποίο ο κύριος ε, ο προσβευτής Ρίτσπερκ απεκάλεσε ατιμορρησία των Ισραηλινών εγκλημάτων αλλά ταυτόχρονα και τις απαντήσεις της ε, Χαμάς ως προς την ανταπόκριση της Χαμάς σε αυτές τις επιθέσεις. Θα ήθελα όμως εγώ να επικεντρωθώ σε ένα θέμα πάνω απ' όλα διότι γνωρίζω ότι όλα τα μέλη της συγκεκριμένη εδώ συνέλευσης έχουν ακούσει πολλά, γνωρίζουν πολλά για την ειρηνευτική διαδικασία. Τόσο πολλά που ομολογώ ότι εκπλήσωμαι για την αθρώα συμμετοχή τους εδώ. Αλλά αυτό αποδεικνύει βέβαια πόσο σημαντική και σοβαρή είναι η κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η δική μας αιμονή στο πάγωμα των ε, επικισμών δεν είναι δική μας προϋπόθεση, είναι δική σας δέσμευση από το φύλλο πορείας. Ταυτόχρονα όμως θα πω και γιατί δεν είναι η μόνη υποχρέωση αυτή, γιατί όμως χωρίς να είναι η μόνη υποχρέωση είναι τόσο σημαντική, διότι και υπό το φως των, διαπραγματεύσεων μας, των ε, εμπειριών μας από τις διαπραγματεύσεις θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι έχει αποδιαρθρωθεί η έννοια κάθε εμπιστοσύνη σε επίπεδο όχι μόνο Παλαιστινιών αλλά γενικά αραβικής κοινή γνώμης και θα σα εξηγήσω τι εννοώ. Η επέκταση των επικισμών έχει ουσιαστικά οδηγήσει στην αναγνώριση αυτής της ειρηνευτικής διαδικασίας ως μόνο φίλος οικής που προσπαθεί να, να ε, καλύψει την συνεχιζόμενη κατάσταση πιέσης επικισμούς όχι μόνο σε επίσημη μορφή αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι παρέχεται κάθε διευκόλυνση για την επιβίωση των επικισμών αυτών. Δηλαδή και διόδη υπάρχουν και δημόσια κτίρια και νοσοκομεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα ανοικοδομούνται και κάθε είδους δημόσιες υποδομές που προσφέρει το Ισραηλινό κράτος στους επικισμούς αυτούς όπως ε, αποχέτευση, ίδρευση, άρδευση, ηλεκτρισμό τηλέφωνο ακόμη. Έτσι λοιπόν, παρά τις όποιες δεσμεύσεις ή προτάσεις της κυβέρνησης του Νετανιάχου να αποζ... κλειστεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ από του αποκλεισμού να αποκλειστούν 3.500 από αυτού που δεν ακολούθησαν. Αυτέ είναι οι του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Είναι ισοδύναμε με το να λέμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα για ειρήνη. Και έχω σημειώσει ότι εσείς ε, κύριε Πρεσβευτή ε, κύριε, κύριε θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει λύση δύο κρατών. Εγώ ύστερα από τρει εβδομάδε πέρασα στην Παλαιστίνη. Δεν βλέπω ακριβώ πού θα μπορούσε να τοποθετηθεί το Παλαιστινιακό κράτο δεδομένη τη ταχύτητα τη επεκτάσεω των επικισμών. Και πάνω απ' όλα αναφέρομαι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι κατεχόμενο έδαφο, το γνωρίζει όλο ο κόσμο και η Αμερικανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπορείτε να την, αποκλείσετε από το πάγωμα των επικισμών λέγοντα ότι θέλετε να δοθεί μια λύση δύο κρατών. Διότι θα πρέπει η Ανατολική Ιερουσαλήμ να είναι η πρωτεύουσα των δύο κρατών. Χωρίς Ανατολική Ιερουσαλήμ δύο κράτη δεν μπορούν να υπάρχουν. Επίσης, οι τρεις ε, θύλακες επικισμών που θέλετε να αποκλείσετε με τις 3.500 νέες μονάδες, πρόταση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, σημαίνουν επέκταση του πληθυσμού της Άριελ, του μεγαλύτερου δηλαδή επικισμού στο βορρά, Μάλια, Μπιλίμ στην ε, στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ και της Ισιών στην ε, ε, περιοχή της Δυτικής Όχθης, ότι με αποτέλεσμα το Παλαιστινιακό κράτος να παραμείνει μόνο ένα κράτος θυλάκων, δηλαδή αποκομμένων κομματιών εδάφους που δεν θα έχουν μεταξύ τους σύνδεση, δηλαδή δεν θα έχουν και καμία βιωσιμότητα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να επιβιώσει ένα τέτοιο κράτος και στην ε, πράξη. Αυτοί οι επικισμοί υποδαβλίζουν οποιαδήποτε πιθανότητα για λύση. Και επίσης Σημειώνω ότι το ζήτημα των επικισμών δεν είναι θέμα ε, προϋποθέσεων. Έχει πρακτικό χαρακτήρα η σημασία ε, που αποδίδεται στους, επικισμούς και γι' αυτό κάθε φορά υπενθυμίζουμε τη δέσμευση της Ισραηλινής κυβέρνησης και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να μιλούμε για λύση δύο κρατών εκτός και, ε, να σταματήσουν οι επικισμοί ή εκτός και αν θέλετε μία λύση ενός κράτους αλλά διεθνοτικού πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε και να συζητήσουμε με διαφορετικούς όνου. Συνεχίζω λέγοντα ότι οι επικισμοί στην Ιερουσαλήμ ισοδυναμούν με 35% της στέγη που ε, ανεγείρεται στο Ισραήλ. Με 45% πληθυσμό των επικιστών στην Δυτική Όχθη σήμερα, 500.000 δηλαδή επικιστές, μισό εκατομμύριο, και επικισμούς που δεν είναι η μόνη πολιτική της νεαράς κυβέρνησης του Νετανιάχου διότι αυτή έχει αναλάβει και επέκταση των ε, επικισμών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στο Σιχρανάχ και στο Σελουέν έχει προχωρήσει σε κατεδάφιση οικειών και επίσης εν τέλει τις τελευταίες εβδομάδες δυστυχώς με πολύ ανησυχητική κίνηση προχώρησαν επικιστές στην περιοχή του Χαράμι Σερίφ. Το επέτρεψαν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Τι ερωτικέ δυνάμει κατοχή. Πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Εγώ ήμουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που συνέβη αυτό. Και λέω ανησυχητικό διότι πραγματικά ε, υπονομεύει, μάλλον ε, κάθε είδου ε, ριζοσπαστισμό θρησκευτικό για το Χαράμι Σερίφ. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ιερό χώρο για κάθε ε, μουσουλμάνο όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους και ταυτόχρονα η κίνηση αυτή μας αποστερεί, αποστελεί τους Παλαιστίνιους από, μια βασική, από ένα βασικό χώρο θρησκείας και λατρείας. Ύστερα από την επίθεση εις βάρος του τεμένους του Αβραάμ, αυτή η στάση σας στην υπόθεση του Χαράμι Σερίφ αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για οποιαδήποτε σχέση ειρήνης ή ειρήνευσης με ολόκληρο τον αραβικό κόσμο και όχι μόνο για την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είπατε, πρέσβη, κύριε Κυριέλ, ότι θέλετε να είναι μέρος της λύσης η Ιερουσαλήμ. Αν δεν το είπατε, ίσως το σκεφτήκατε. Ναι, αλλά είναι και κομμάτι του κράτους. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τους πρόσφυγες, τις επικισμούς, τα σύνορα, τους δατίνους πόρους να αναγνωρίσετε ότι αυτό θα είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που θα χρειαστεί να συζητήσουμε ως προς το καθεστώς ε, του όποιου κράτους. Αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν χωρίς να προκαθοριστεί με τέτοιου είδους ε, κινήσεις τελεσμένων το μελλοντικό καθεστώς της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Εμείς δεν ε, προσπαθούμε να απαλλαγούμε από τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας. Όπως είπα, εμείς η Παλαιστινιακή Αρχή τα τελευταία 18 χρόνια και με τον Πρόεδρο Αραφάτ και με τον Πρόεδρο Αμπάς αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες μας παρά το γεγονός ότι τελούμε υποκατοχή και θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο Ισραηλοπαλαιστινιακή ε, ευθύνη ή καθήκον των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων αλλά ολόκληρη τη ε, διεθνού κοινότητα να επιβάλλουν την ε, ορθή εφαρμογή των κανόνων του διεθνού δικαίου. Και θα πρέπει και οι Ισραηλοί να γνωρίσουν την εφαρμογή των διεθνών του διεθνού δικαίου όπω κάθε κράτο μέλο των Ηνωμένων Εθνών όπως και όλων των εδώ εκπροσωπουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των αραβικών κρατών. Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι προκειμένου να προχωρήσουμε χρειαζόμαστε καλύτερη προστασία του τεχνικού δελτίου ή των όρων των όσων πράττουμε. Ο πρόεδρος Ομπάμα με την ε, τοποθέτησή του, όχι μόνο για την Παλαιστινιακή, για, την, ε, για το Μεσανατολικό, την ειρηνευτική διαδικασία στη Μεσανατολία, αλλά γενικά με την τοποθέτησή του έχει γεννήσει τεράστιες ελπίδες για ειρήνη, ύστερα από δύο ε, θητείες προέδρου, δύο ε, αλλεπάλληλες προεδρικές θητείες, οι οποίες μόνο πόλεμο και καταστροφές έφεραν στον κόσμο. Αυτή η ελπίδα λοιπόν για την ειρήνη που γέννησε και η διακήρυξη του ίδιου του Προέδρου Ομπάμα ότι θα στηρίξει την ε, εξωτερική του πολιτική στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου με το κλείσιμο αφενός του, ε, του Γουαντάναμο αλλά και της ε, προσφοράς για έναρξη διαπραγματεύσεων του όλους τους εταίρους συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του Ιράν αποτελούν για μας μεγάλη πηγή ελπίδας. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Παρά την κατοχή εμείς αποφασίσαμε και προσπαθούμε να ανοικοδομήσουμε υποδομές για το κράτος μας. Και ελπίζουμε και με τη δική μας σας βοήθεια τα επόμενα δύο χρόνια και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστώ την Προεδρία η οποία είπε τόσα θετικά πράγματα για το διετές μας πρόγραμμα για την πρόταση δηλαδή για περάτωση της κατοχής και την ανάπτυξη κράτους γιατί βέβαια προφανώς ο κύριος εταίρος μας, ο ένας από τους κύριους εταίρους μας θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη τόσο γενναιόδορη προσφορά της. Πλην όμως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ανοικοδομήσουμε κράτος με όλη τη γενοδορία των χορηγών μας, Αράβων, Αμερικανών ή Ευρωπαίων εάν δεν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάσταση όπου θα έχει περατωθεί η κατοχή και αν δεν συνεχίσουμε τον αγώνα για την ένωση, σκληρό αγώνα για την ένωση των πολιτικών κινημάτων για τους ε, Παλαιστινίους υπό την, υπό την οργάνωση για την ε, απελευθέρωση Παλαιστίνης και σε συνεργασία μέσα στον ε, διάλογο της Χαμάς και της Φατάχ. Με τις προσπάθειες που μας έχουν, στις οποίες μας έχουν στηρίξει οι φίλοι μας ε, στον δρόμο για την επιτυχία και θα ήθελα να πω ότι ο μόνος τρόπος να κριθεί το ποιος εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους είναι οι δημοκρατικές εκλογές. Αυτό με βάση και τις προτάσεις της Αιγυπτιακής κυβέρνησης πρέπει να λάβει χώρα τον Ιανουάριο ή μη το αργότερο έως τον Ιούνιο και πάντως ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να περιμένουμε τέτοιου είδου εκλογική αναμάκρυση προκειμένου να μπορέσουμε και σε συνεργασία με του εταίρου και ελπίζω όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τι Ηνωμένε Πολιτείε να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη και τι εγγύσει που χρειάζονται οι Παλαιστίνοι προκειμένου να ανακτήσουν εμπιστοσύνη σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία που, που το τελευταίο καιρό έχει χάσει την αξιοπιστία τη. Ευχαριστώ τη Γενική Εκπρόσωπο. Πριν περάσουμε στις παρεμβάσεις σας, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κέρτιν. Όταν σα παρουσίασα, κυρία Κέρτιν, προηγουμένω δεν είχατε ακόμα φτάσει. Θα θέλαμε να ακούσουμε ποιε είναι οι αμερικανικέ προσπάθειε για την ειρήνη, τη στιγμή που η Χίλαρη Κλίντον έκανε αυτή την γρήγορη επίσκεψη στη Μέση Ανατολή και όπου χθε στο Μαρόκο συναντήθηκε με του υπουργού εξωτερικών των αραβικών χωρών. Είσαστε υφυπουργό πολιτικών υποθέσεων και σύμβουλο για την Μέση Ανατολή στην Αμερικανική Αποστολή στι Ηνωμένε Πολιτείε, στην Αμερικανική Αντιπροσωπεία στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ και καλημέρα. Φυσικά θα μιλήσω αγγλικά. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι μπροστά σα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που με κάλεσε, που κάλεσε την, Αμερικανική πλευρά στη συνάντηση αυτή. Στην, εγώ είχα βάσει κέντρα την Τινησία για τέσσερα χρόνια ε, και αναγνωρίζω διάφορα πρόσωπα από την Τινησία καθώς και από την πρεσβεία ε, της Αιγύπτου, στην Αίγυπτο μάλλον. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να μιλήσουμε για τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των χωρών μας, των πολιτισμών μας, ε, των περιφερειών μας και να μιλήσουμε για τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν και που καταβάλλονται για να προχωρήσει η ειρήνη και η σταθερότητα όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τελικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι οτιδήποτε συμβεί σε μια περιοχή του κόσμου επηρεάζει πάρα πολύ άλλες περιοχές του κόσμου. Νομίζω λοιπόν, κάτι που ίσως ξέρετε, ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, βρίσκεται σήμερα και αύριο στη Ουάσιγκτον για μια σύνοδο κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Ηνωμένων Πολιτειών που συνήθω γίνεται κάθε χρόνο και αυτή είναι η πρώτη επίσημη σύνοδο κορυφή ε, με τη νέα κυβέρνηση Ομπάμα. Έγινε την άνοιξη στην Πράγα μια ανεπίσημη σύνοδο κορυφή. Αυτή είναι η επίσημη σύνοδο κορυφή. Και μεταξύ των θεμάτων στη μερίσια διάταξη για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο με την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά θα είναι οι προσπάθειε για να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να ανοίξουν και να αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Όχι απλώς να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά να έχουν και ένα στόχο να υπάρξει συμφωνία όπου τα δύο κράτη θα ζουν ε, δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια. Οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών θα μιλήσουν επίσης για το Αφγανιστάν, για την κλιματική αλλαγή, για οικονομικά θέματα μια σειρά θεμάτων που μας ενδιαφέρουν από κοινό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στη Ουάσιγκτον, η Υπουργό Εξωτερικών Χίλαρη Κλίντον, αυτή τη στιγμή νομίζω, εκφωνεί μια ομιλία στο Φόρουμ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο Μαρακέ στο Μαρόκο. Η ομιλία της έχει προετοιμαστεί εδώ και καιρό Και φυσικά αυτή τη στιγμή εκφωνεί το λόγο της, δεν μπορώ φυσικά να σας πω τι ακριβώς λέει, αλλά ο στόχος της ομιλίας ήταν να αναγγείλει διάφορες πρωτοβουλίες που οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα προωθήσουν στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής για να υπάρξει εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών, ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν διάφορα θέματα που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά, όπως παραδείγματο χάρη η πρόοδος ε, των γυναικών ε, και συμμετοχή τους ε, στην πολιτική, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία δεσμών μέσω πολιτιστικών προγραμμάτων μεταξύ των λαών μας. Αυτή είναι μια ομιλία που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Επίσης, όταν έφτασε στο Μαρόκο, είχε διάφορες επαφές και συναντήσεις με την ηγεσία διαφόρων χωρών της Μέσης Ανατολής, καθώς και με την ηγεσία του Αραβικού Συνδέσμου για να μιλήσει για τις προσπάθειές μας, τις κοινέ προσπάθειές μας για να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εξαιτίας των ανησυχιών που έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες, σκοπεύει η κυρία Κλίντον να πάει στο Κάιρο για να συνεχίσει αυτές τις συζητήσεις. Αυτή η θέληση σε μια φορτωμένη χρονική στιγμή να σταματήσει σε αυτό το θέμα, τη στιγμή που συναντάει την ηγεσία παραδείγματο χάρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. παρόλα αυτά θα πάει στο Κάιρο για να συνεχιστούν οι συζητήσει για το πώ θα βοηθήσουμε του Ιτζαηλινού και του Παλαιστίνιου να ξαναρχίσουν τι διαπραγματεύσει. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά ένα δείχτης, ένα σημάδι ε, τη σημασία που δίνει ο πρόεδρο Ομπάμα στο θέμα αυτό. Όπως υπόθηκε ήδη, και από την εκπρόσωπο της Παλαιστίνης, ο πρόεδρος Ομπάμα ξεκαθάρισε τη δέσμευσή του να υπάρξει ε, ειρήνη στην Μέση Ανατολή όταν διόρισε τον Τζορτζ Μίτζελ ειδικό απεσταλμένο τη Μέση Ανατολή από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του. Ε, ο κύριος Μίτζελ είναι ένας πεπειραμένος άνθρωπος. Εγώ είμαι Αμερικανίδα Ιρλανδικής καταγωγής και γνωρίζω τι προσπάθειες έχουν γίνει για να βοηθήσουμε τους Ιρλανδούς να κάνουν κάποιους πολύ σοβαρούς συμβιβασμούς που οδήγησαν στην ειρήνη και στην ευημερία πριν από 10 χρόνια. Που πριν 10 χρόνια μάλλον θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί. Ο κύριος Μίτσελ από τον Ιανουάριο δούλεψε ακαταπώνητα για να βρει έναν τρόπο να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Ισραηλινού και του ε, Παλαιστίνου με σκοπό να δημιουργηθούν δύο κράτη που θα ζουν δίπλα-δίπλα. Θα θέλαμε το Ισραήλ να είναι ασφαλέ και η Παλαιστίνη να είναι ένα συνεχέ κράτο που θα ζει με ασφάλεια. Ε, η κατοχή ξεκίνησε το 1967 θα θέλαμε να σταματήσει τώρα. Ο πρόεδρος Ομπάμα ξεκαθάρισε πολλές φορές ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα θέματα του μόνιμου καθεστώτος, ε, σύνορα, ασφάλεια, ε, πρόσφυγες. Είναι ένας δύσκολος δρόμος και μερικές φορές όπως σήμερα και με τις ανταλλαγές που έγιναν το Σαββατοκύριακο ε, μοιάζει δύσκολο να μπορεί να υλοποιηθεί. Αλλά ο πρόεδρος και η Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος Μίτσελ ο γερουσιαστής κ. Μίσελ είναι και οι άνθρωποι βεβαίως της περιοχής είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό. Σήμερα ε, εστιάσαμε σε αυτές τις προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να μιλήσω ε, και για άλλες ε, προτεραιότητες της ε, κυβέρνησης γιατί συνδέονται με τους βασικούς μας στόχους. Πέρα από την ενθάρρυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης θα θέλαμε ε, να υπάρχει ευρύτερη ειρήνη στην ε, περιοχή μεταξύ ε, Ισραήλ και Συρίας και Ισραήλ και Λιβάνου. Μετά το παράδειγμα που έδωσαν η, η Αίγυπτος και η, η Ορδανία με τις ειρηνευτικές συμφωνίες πριν από πολλά χρόνια. Επίσης, ε, μια άλλη δέσμευση είναι ο μη πολλαπλασιασμός των ε, πυρηνικών. Αυτό νομίζω θα εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Θέλουμε να παρεμποδίσουμε ε, τον πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων, τον τρόπο εξάπλωσή του. Θα πρέπει οι έξι ε, πυρηνικέ δυνάμει ε, να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά του όπλα για ειρηνικού σκοπού. Οι έξι πυρηνικέ δυνάμει περιοχή. Αυτό το είπε ο πρόεδρο Ομπάμα στην Πράγα ε, όταν μίλησε ε, για τις προσπάθειες που κάνουμε και εμείς μαζί με τους Ρώσους για να μειώσουμε τα, τα πυρηνικά, κάτι που είναι βασική προτεραιότητα της ε, κυβέρνησης. Όπως ο πρόεδρος είπε στην ομιλία του στο Κάιρο, θα θέλαμε να υπάρχουν ε, εταιρικέ σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής που υποστηρίζει τους στόχους για τους οποίους θα μιλήσει η Χίλαρη Κλίντον. εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και υγεία. Θα θέλαμε να δουλέψουμε με τους κατοίκους της περιοχής για να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσωπευτικότητα, ε, συμμετοχή, ε, σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών και των θρησκευτικών μειονοτήτων. Ε, ένας από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης αυτής είναι η έμφαση στο διάλογο. Η κυβέρνηση και ο πρόεδρος ειδικά ανέλαβαν τα καθήκοντά τους πιστεύοντας ότι το να μην συνδιαλέγεσαι με τις άλλες χώρες δεν οδηγεί πουθενά. Όπως ξέρετε έχουμε ξεκινήσει διαλόγους με τους εταίρους μας ε, στην διαδικασία P5 1 για να ξεκινήσουμε το διάλογο με το Ιράν, ούτω ώστε να αποφύγουμε να απειλεί όλη την περιοχή με την ε, εξασφάλιση πυρηνικών όπλων. Και τώρα, ε, αφού κάναμε αυτή την κίνηση, περιμένουμε απάντηση από το Ιράν σε μια συγκεκριμένη πρόταση, ούτω ώστε να Ε, το εμπλουτισμένο ουράνιο να χρησιμοποιηθεί μόνο για επιστημονικούς σκοπούς. Ε, αυτή είναι η προσφορά που κάναμε και ελπίζουμε να το δεχθεί το Ιράν. Δεν τελειώνουν αυτά τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια κίνηση και μια απόδειξη των θετικών επιπτώσεων του διαλόγου. Επίσης έχουμε ανοιχτό διάλογο με τη Συρία. Πιστεύουμε ότι η Συρία και η ΕΠΑ έχουν κοινά, κάποια κοινά συμφέροντα, παραδείγματο χάρη ευρεία ειρήνη στην περιοχή και ότι η Συρία θα μπορούσε δυνητικά να παίξει επικοδομητικό ρόλο για να υλοποιηθούν οι κοινοί μα στόχοι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ζητήσει από τη Συρία να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα που μα ανησυχούν. Επίση, ο πρόεδρο έχει λάβει μέτρα για να υλοποιήσει την δέσμευση που έδωσε προεκλογικά να, για να φύγουν τα στατεύματά μας από το Ιράκ. Ε, φυσικά υπάρχουν ακόμα σημάδια βίας και υπάρχουν ε, προκλήσεις για την ε, κυβέρνηση του Ιράκ και τον Ιρακινό λαό. Εμείς θα βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Ιράκ, αλλά νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει. Κάποιοι άλλοι ανέφεραν τη δέσμευση του Ιράκ να κλείσει το, τη φυλακή του Γκουαντάναμο. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Είναι ένα πρόγραμμα που κληρονομήσαμε την προηγούμενη κυβέρνηση και ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί να το κλείσει μέσα σε έναν χρόνο. Ίσως μπορεί να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα, αλλά θεωρεί ότι είναι βασική προτεραιότητα και ο Υπουργό Εξωτερικών και ο Υπουργό Δικαιοσύνη ε, κάνουν ό,τι μπορούν για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Επίση, υπάρχουν και διάφορε άλλε προκλήσει στην περιοχή και πιστεύουμε ότι συνδέονται μεταξύ τους. Επίσης όμως πιστεύουμε ότι το θέμα το οποίο συζητήσαμε περισσότερο σήμερα το πρωί, δηλαδή η σημασία της επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και, της, και των Παλαιστινίων για να τελεσφορήσει ο ε, στόχο των δύο κρατών είναι βασική προτεραιότητα αυτή τη κυβέρνηση. Και αυτό δείχνουν και οι αποφάσει και οι προσπάθειε που καταβάλει και ο πρόεδρο, η υπουργό εξωτερικών, ο γερουσιαστή Μίτσελ δείχνουμε τη θέλησή μας να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ούτω ώστε να ξεκινήσει ξανά η όλη διαδικασία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνε του. Ε, δεν έχουμε τέτοιε αυταπάτε. Πιστεύουμε ότι κάθε χώρα που εκπροσωπείται εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, οι διάφοροι ε, περιφερειακοί ηγέτε, ε, όπω η Αίγυπτος, είναι κράτη κλειδιά της διαδικασίας και αυτή η προσπάθεια απαιτεί και συμβιβασμό και επιμονή από όλους μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται σε αυτό το στόχο και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους ε, της περιοχής για να τον πετύχουμε. Σας ευχαριστώ και περιμένω να ακούσω και τις ερωτήσεις σας. Ε. Ευχαριστούμε πολύ. Η τελευταία συνεδρίαση του Προεδρείου του 4η Ιουλίου ήταν μια συνεδρίαση όπου πρότεινα αντιπροσωπεία τη συνέλευσή μα να πάει στη Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με μέλη του Κογκρέσου, τουλάχιστον με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ενδεχομένω, αν είναι δυνατόν, και με την Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Κλίντον. Θα αποφασίσουμε στο Προεδρείο της 20 Νοεμβρίου ακριβώς πώς θα οργανώσουμε αυτή την επίσκεψη. Τώρα, Ξεκινάει η συζήτηση. Θα ήθελα να αποφύγουμε μόνο λόγους και μακρηγορήσεις. Καλό θα ήταν να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Εσυσλή πρώτα από την Αιγυπτιακή Αντιπροσωπεία, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Στο όνομα του Πολυέλου και Συνεχού Θεού θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς, Πρόεδρε, και όλους τους παρόντες εδώ. Θέλω να πω ευθύ εξ αρχής ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μια περιοχή όπου είχαμε πολλές θετικές εξελίξεις τον τελευταίο καιρό όσον αφορά το Παλαιστινιακό έγιναν πολλές προσπάθειες από διάφορες πλευρές προκειμένου να πετύχουμε μια συνολική και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Έτσι λοιπόν το Παλαιστινιακό πέρασε από διάφορα στάδια. Είχαμε και οπισθοχωρήσεις μετά την επίθεση στη Γάζα του Ισραήλ. Η επίθεση αυτή τάραξε τις συνειδήσεις όλου του κόσμου. Και αυτό εξαιτίας ε, των χιλιάδων νεκρών που είχαμε μετά την επίθεση αυτή. Και τώρα τι γίνεται, στάξαμε στην, ε, στο Ιεροσόλυμα, σαμποτάρεται η περιοχή αυτή. Και εμποδίζονται οι πιστοί που θέλουν να πάνε εκεί να προσευχηθούν. Αυτό σημαίνει, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι η επίθεση της Γάζας οδήγησε στην αποτυχία της επίτευξης οποιοδήποτε πολιτικού στόχου. Δεν οδήγησε στο να μειωθεί η αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού, ούτε μείωσε την επιθυμία των ε, Παλαιστινίων να έχουν ελευθερία στην περιοχή τους δεν οδήγησε ούτε και σε καρποφόρα αποτελέσματα προκειμένου να έχουμε μια δίκαια και βιώσιμη λύση για το Παλαιστινιακό, παρά τις προσπάθειες που έκανε η Αίγυπτος προς αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έρθουν όλα τα εμπόδια που παραμένουν όσον αφορά την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου είπε ότι οι απαιτήσει του Ισραήλ, προκειμένου το Ισραήλ να είναι ένα εθνικό κράτος για τους Εβραίους, απειλεί τη βιωσιμότητα της ειρήνης. Και κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο έτοιμο στη διεκδίκηση αυτή, ούτε στη Μέση Ανατολή, ούτε και πουθενά αλλού. Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε υπόψη μα ότι για να πετύχουμε μια βιώσιμη και δίκαια ειρήνη πρέπει να έχουμε και συμμετοχή όλων των πλευρών και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει βούληση εφαρμογής των συμφωνιών προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η βούληση της διεθνούς κοινότητας πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και αυτό προς το συμφέρον του Παλαιστινιακού λαού. Ο εξοχότης του πρέσβης είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε ειρήνη χωρίς διαπραγματεύσεις. Και εγώ θα έλεγα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις χωρίς να ε, ξεκινήσουμε με τους επικισμούς. Και αυτό είναι που η Παλαιστίνια πρέσβης μόλις δήλωσε και αυτό έχει πει και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, ο Μαχμούτα Μπάς. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε, ότι η επιτυχία των προσπαθειών της Αιγύπτου προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορές στην περιοχή και να πετύχουμε μια δίκαια και συνολική ειρήνη υπέρ των δύο κρατών σημαίνει πρώτα απ' όλα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, η συμμόρφωση του Ισραήλ στις προϋποθέσεις που βάζει η διεθνής κοινότητα. Μεταξύ άλλων και τελευταία, η αύξηση του ρυθμού οικοδόμησης επικισμών στη Δυτική Όχθη είναι πάρα πολύ σημαντικό η διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί και να πείσει το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην περιοχή. Επίσης, από την άλλη μεριά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και εθνική ενότητα μεταξύ των Παλαιστινίων και να πιστούν, να, πιστούν, να είναι ενωμένοι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνία συμφιλίωσης. Μόνο έτσι θα στηριχθούν καλά οι διαπραγματεύσεις. Ακούσαμε τις δηλώσεις για την δέσμευση να υπάρξει ένα Παλαιστινιακό κράτος με τους τόπους να είναι βιώσιμο κλπ. Έχουμε ακούσει πολλές δεσμεύσεις. οι κινήσεις που γίνονται, οι δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών ε, Κλίντον στην σημερινή συγκυρία, οι συναντήσεις που έχει με τους Υπουργούς Εξωτερικών ε, των Αραβικών χωρών ε, στο Μαρόκο αποτελούν παράδειγμα των συνεχών προσπαθειών που γίνονται και ευχαρίστω να την υποδεχτούμε και πάλι στο Κάιρο για να συνεχίσει τις προσπάθειές της. Θα συναντηθεί με πολλές πλευρές από τον Αιγυπτιακό λαό. Θα την δεχτούμε ευχαρίστως και πάλι στο Κάιρο, όπως ε, και ο πρόεδρος. Εκεί είχαμε και μια ιστορική ομιλία που έδωσε ελπίδες καινούργιες για την ειρηνευτική διαδικασία. Ιδίως μετά από την ε, έλευση του νέου πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι βασικά που οδήγησε τον κόσμο σε νέες ελπίδες για ειρήνη στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βέγκελ τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Εδώ μιλούμε για ειρήνη και πόλεμο μέσα και γύρω από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Προφανώς τα ίδια αυτά προβλήματα θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε και στο πλαίσιο ιουδήποτε άλλου θέματος, ζητήματος, περιφερειακής πρωτοβουλίας ή οργανώσεως διότι αποτελούν τη ρίζα κάθε άλλης κρίσεως μέσα και γύρω από την Ευρώπη. Δεν είναι ένα τοπικού χαρακτήρα πρόβλημα, είναι ένα παγκόσμιο χαρακτήρα πρόβλημα, παλαιό πρόβλημα που έχει διαρκώς επεκτάσεις και, και διακλαδώσεις και γεννά κινδύνους πολέμων και δεινών σε όλο τον κόσμο. τη χάνει να επιστρέφω από την ε, Ιορδανία μου και την προηγούμενη εβδομάδα όπου συναντήθηκα με αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται και με ανθρωπιστική βοήθεια για την Παλαιστίνη και αμφισβητώ τα όσα είπε ο πρεσβευτής Κουριέλα ότι είναι ανοιχτή, δηλαδή, ανοιχτά οι δίωδοι της ανθρωπιστικής βοήθειας ή οι θύρες ανθρωπιστικής βοήθειας. Εγώ μόνο για κλειστές θύρες άκουσα να γίνεται λόγος. Και όσο ήμουν εκεί, στις εφημερίδες και στον τύπο διάβαζα εκθέσει τη Διεθνούς Αμνηστίας ως προς τα προβλήματα στην ίδρυυση. Και δεν είναι δύσκολο στην περιοχή να αντιληφθεί κανείς πόσο τεράστιο είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας. Είναι παρόν παντού. Φυσικά μπορεί κανείς να συζητεί για την, ε, τα σχέδια περί εκτροπής ε, του ε, Ιορδάνη ποταμού ή για την ξηρασία ή τη λειψιδρία που μπορεί να γεννά αυτή σε άλλες περιοχές, περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον τα εδάφη του Παλαιστινιακού κράτους. Θα μπορούσαν να είναι στο μέλλον το Παλαιστινιακό κράτος. Και αυτό το οποίο με ε, συγκλώνησε περισσότερο σήμερα ήταν η χρήση του όρου τρομοκρατική οντότης. Εγώ, κύριε Πρεσβευτάκη, ήμουν πρεσβευτή ο ίδιος για πολλά χρόνια. Θα σας πω ότι χρησιμοποιήσετε όρο τον οποίο δεν θα έπρεπε να βάλετε στο σώμα σας και οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη από το λαό της Γάζας, από τα παιδιά, από τους ηλικιωμένου, από όλους όσοι υπέφεραν λόγω πράξεων άδικων πολιτικής επιλογής λόγω της αποτυχίας της κάθε πλευράς να εξεύρει το στο πρόβλημα και εκείνοι οι οποίοι έχουν την, ε, το μικρότερο μερίδιο της ευθύνης που είναι οι αθώοι είναι εκείνοι οι οποίοι υπέφεραν το περισσότερο στη λόρδα της Γάζας. Δεν είναι τρομοκράτες. Είναι απλώς οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από τα δεινά αυτά. Και πρόεδρε, ακολουθώντας τη συμβουλή σας δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα απλώς να διατυπώσω κάποιες παρατηρήσεις. Μιλούμε για πολιτική επίδραση, αντίκτυπο της κρίσης στην περιοχή. Αλλά εγώ περισσότερο θα ήθελα να μιλήσω για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ορδά της Σήμερα ήρθα με καθυστέρηση στη συνεδρίαση ε, λόγω της κακοκαιρίας στη Λουμπλιάνα. Άρχισε ο χειμώνας, είχαμε χιονοθύελα. Και άκουσα εγώ όσο ήμουν στην Ορδανία να λένε όλοι ο χειμώνας αυτός θα είναι ε, πολύ δρυμής και για την Λόριδα της Γάζας. Χρειάζεται λοιπόν ανθρωπιστική βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει τώρα. Ιδιαίτερη έμφαση λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε στην ανθρωπιστική κατάσταση σήμερα στη Λόριδα της Γάζας και να δούμε, να εξετάσουμε εάν όντως μπορούν ε, απρόσκοπτα να προχωρήσουν ε, τα ε, φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια ή εάν έχουν σταματήσει κάπου στο δρόμο και γιατί. Να σας εμπιστευτώ όταν μου λέτε ότι είναι ανοιχτέ οι δύο δι, αλλά θα εμπιστευτώ και εκείνους στην Ιορδανία που καθημερινά ασχολούνται με την ε, μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό ήταν το πρώτο που θέλω να πω. Και δεύτερον, βλέπω με ικανοποίηση εδώ παρουσία των εκπροσώπων όλων των κρατών που ενδιαφέρονται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι καλό το ότι προσπαθείτε να είστε επικοδομητικοί, ευχάριστοι μερικές φορές ο ένας τον άλλον. Αλλά, και ύστερα από τόσα είπε και ο ε, πρέσβης ε, ε, της Αιγύπτου και όσα επίσης ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το τέμενος Αλαξά, δεν έχω παρά να πω ότι ήταν μια σκληρή ε, ανετίαστη πρόκληση και άκουσα τον κύριο Κλίντον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ που μίλησε στη Λουμπλιάνα πρόσφατα για άλλη μία απόπειρα να προκληθούν προβλήματα γύρω από το τέμενος Σαλαξά και θυμάστε ότι ήταν ε, η επίσκεψη του Σαρών εκεί. Εκείνος ουσιαστικά προκάλεσε ε, ε, το ξέσπασμα ανυπέρβλητων δυσκολιών και προβλημάτων μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών ή αλλιώς μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων. Δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο και πρέπει εμείς να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των μουσουλμάνων σε ένα ιερό για αυτούς τόπο λατρείας. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί κανείς να τους προκαλεί. Δεν μπορεί κανείς να προσπαθεί να τους ταπεινώσει. Αυτό είναι άλλο ένα σημείο στο οποίο ήθελα να αναφερθώ και ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ελπίζοντας ότι δεν καταχράστην του χρόνου. Ευχαριστώ. Ο πρέσβης κύριος Κιουριέλ θα σας απαντήσει, αλλά θα ήθελα πρώτα να ακούσω διάφορες ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Όλοι έχετε σημειωθεί, όλοι όσοι έχετε σηκώσει το χέρι. Έχουμε ένα πλήρη κατάλογο, όλοι θα πάρετε το λόγο, μην ανησυχείτε. Ανησυχείτε, ξέρουμε, έχουμε καταγράψει τα ονόματά σας. Άλλο καθένας με τη σειρά του. Ο κύριος Σαντούκα. Σας παρακαλώ με συντομία και λακωνικότητα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους κύριους συμμιλητές και θα ήθελα καταρχάς να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτά που ακούσαμε από τους κύριους ομιλητές. Θα κάνω κάποια σχόλια καταρχάς στα όσα είπε ο Ισραηλινός πρέσβης, ο κύριος Κουριέλα. Ο πρέσβης επιβεβαίωσε την σημασία της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Άκουσα κάποια θετικά πράγματα που με χαροποίησαν επίσης από την κυρία Κέρτιν, η οποία είπε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να υπάρξει ειρήνη και να δημιουργηθούν δύο κράτη στην περιοχή. Τελικά. Πιστεύουμε ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαμε με τους ε, Ισραηλινούς ε, εταίρους μας ήταν διαπραγματεύσεις για τις διαπραγματεύσεις. Ο στόχος δεν ήταν να υπάρξει τελικά ειρήνη και μια δικρατική λύση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την εντύπωση δίνουν οι Ισραηλινοί εταίροι μας από τις μέχρι τούδε διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Χαξαμίρ ο πρώην ε, Πρωθυπουργό του Ισραήλ είπε στην αρχή των διαπραγματεύσεων ότι ήλπιζε να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις για 10 χρόνια ή και ατέρμονα. Αυτό το είπε στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό να πω ότι συμπεράναμε από πλευράς Παλαιστινίων ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθούσε απλώς να πετύχει τι, το να διαπραγματευτεί και μόνο. Και όχι να οδηγήσουν κάπου διαπραγματεύσεις, δηλαδή να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή μας και να δημιουργηθούν δύο κράτη, ένα για το Ισραήλ και ένα για την Παλαιστίνη. Όπω είπε ο πρέσβης στην ομιλία του, αυτή η δικρατική λύση ε, υπάρχει ήδη από τη δήλωση του 1947. Όλες οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με την Ισραηλινή κυβέρνηση στην πραγματικότητα τέλειωσαν πώς ε, με το να παίρνει τη σκητάλη νέα κυβέρνηση από την παλιά και εμείς να ζητάμε από κάθε νέα κυβέρνηση να ξαναρχίσει τι διαπραγματεύσει γιατί κάθε κυβέρνηση ποτέ δεν σεβόταν τα όσα είχε προσυπογράψει και στα όσα είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει τι. Πρέπει να κοιτάξετε το αρχείο όλων των συμφωνιών που υπογράψαμε για να δείτε πραγματικά του λόγου μου το αληθέ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο πρεσβευτή. <coughs> αναφέρθηκε στην έξοδο από τη Γάζα και στην διάλυση των επικισμών. Ε, είπε ότι το Ισραήλ έφυγε από τη Γάζα και διέλυσε τους επικισμούς, αλλά εξεπλάγησαν οι Ισραηλινοί ε, από τα κακά αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα έγινε ανακατανομή του Ισραηλινού λαού, του Ισραηλινού συγγνώμη στρατού. Και η Γάζα αυτή τη στιγμή είναι μια πολιορκούμενη περιοχή. και τα θαλάσσια σύνορα, τα θαλάσσια περάσματα, καθώς και τα χερσαία περάσματα είναι στα χέρια των Ισραηλινών. Τα κλείνουν και τα ανοίγουν όποτε το επιθυμούν. Και αυτό αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν φύγατε από τη Γάζα και ότι συνεχίζεται η πολιορκία της Λόιδας της Γάζας. Απλώς έχετε ανακατανείμει το στρατό σας στα σύνορα της Γάζας. Δεν απελευθερώσατε τη Γάζα. Η Γάζα δεν έχει απελευθερωθεί. Η Γάζα τελεί υπό Ισραηλινή κατοχή. Υπάρχουν εκεί και Ισραηλινοί πύραυλοι και Ισραηλινά τάγκς και όποτε επιθυμούν να εισβάλλουν πιο βαθιά στη Γάζα, το κάνουν. Δεν θέλω να μιλήσω για τα εγκλήματα που έγιναν στη Γάζα, γιατί η έκθεση Goldstone τα αναφέρει με μεγάλη επάρκεια και ακρίβεια. Ο πρέσβη επίσης ανέφερε ότι πιστεύει στη λύση των δύο κρατών στην περιοχή. Υπάρχει και ένα ρητό που λέει ότι τα έργα είναι καλύτερα από τα λόγια. Αυτό ισχύει και για σας, αγαπητοί. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα Παλαιστινιακό κράτος, αν το επιθυμείτε πραγματικά, τότε τίθεται το εξής ερώτημα. Πώς γίνεται να απαλωτριώνονται γέες, πώς γίνονται να επεκτείνονται οι επικισμοί, πώς γίνεται να φέρνετε μετανάστες απ' έξω που δεν έχουν καμία σχέση με την Παλαιστίνη και, τη Μέση Ανατολή, να τους φέρνετε και τους ε, εγκαθιδρύετε στις ε, περιοχές αυτές διώχνετε τους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους, τα καταστρέφετε, κατάσχεται τη γη τους, κατάσχεται τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Δημιουργήσατε ένα τείχος επίσης στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και περιβάλλει ε, Παλαιστινιακές πόλεις και χωριά. Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότε δεν μπορούν να φτάσουν στι εκμεταλλεύσει του. Οι φοιτητέ δεν μπορούν να φτάσουν στα σχολεία του ε, και στα πανεπιστήμια του. Οι αγρότε δεν μπορούν καν να μαζέψουν τη σοδιά του. Γιατί αυτό το τείχο του παρεμποδίζει στην καθημερινή του μετακίνηση. Οι παράνομοι έπικοι στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν τη γη όπως τους αρέσει. Παρεμποδίζουν τους Παλαιστίνιους αγρότες να φτάσουν στις ελιές τους, να μαζέψουν τη σοδιά τους. Μιλάμε για αυτό το ευλογημένο δέντρο το οποίο, στο οποίο στηρίζονται οι Παλαιστίνοι για να επιβιώσουν, την ελιά. Επίσης ανοίγεται παράπλευρους δρόμους για να συνδέεται τους επικισμούς μεταξύ τους. Εμείς δεν μπορούμε να μαζέψουμε τη σοδιά μας. Εσείς κόβετε τα δέντρα μας, καταστρέφετε την υποδομή μας. Αυτές οι πράξεις βοηθούν για να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος. Προωθούν αυτή τη λύση. Δημιουργείται 600 περίπου φυλάκια. Δημιουργήσατε τα τελευταία χρόνια. Αυτό βοηθάει την Παλαιστινιακή οικονομία βοηθάει τους Παλαιστινίους και τα παλαιστινιακά αγαθά να κινηθούν ελεύθερα. Επίσης βοηθάει την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους κάτι τέτοιο. Επίσης τι κάνετε στην Αραβική Ιερουσαλήμ. Πέστε μου τι κάνατε. Γιατί αλλοιώσατε τη φύση της και την περιβάλλατε από επικισμούς παντού. Γύρω-γύρω υπάρχουν επικισμοί. οι Παλαιστίνοι πολίτες στην Ιερουσαλήμ ή στην ε, Δυτική Γάζα, τι κάνουν, πώς μπορούν να κινηθούν, πώς μπορούν να επισκεφθούν ένα τον άλλον. Τους έχετε απομονώσει. Και η Ιερουσαλήμ τι κέρδισε από τις καταστροφικές σας πολιτικές. Γιατί ο λαός της Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να συμμετάσχει στις οικογενειακές ε, γιορτές. Γιατί το ένα μέλος δεν μπορεί να φτάσει στο άλλο μέλος. Δεν μπορεί να γίνουν επισκέψεις. Έχετε καταστρέψει και τη Δυτική Όχθη και τη Λόριδα της Γάζας. Όλη την υποδομή που υπήρχε. Οι Παλαιστίνοι βουλευτές, οι οποίοι εξελέγησαν σε ελεύθερες εκλογές, που εσείς οι ίδιοι και ο υπόλοιπο κόσμος είπατε ότι είναι ελεύθερες εκλογές, γιατί απάγονται. Γιατί εκδιώκονται από την γη τους, οι οποίοι είναι κατεχόμενοι βέβαια. Και γιατί μεταφέρονται στι φυλακές σας οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί το Ισραήλ κρατάει στις ε, φυλακές του 11.000 ή και παραπάνω Παλαιστίνιους. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση των Παλαιστινίων πολιτών ή των Παλαιστινίων οικογενειών που χάνουν τους συγγενείς τους. Αυτές οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί εμποδίζεται 11.000 άτομα που είναι φυλακισμένοι από το να δουλέψουν. Και δεν μπορούν να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Η πρόεδρος μου κάνει νόημα να ολοκληρώσω. Θα ήθελα να πάω τώρα σε ένα βασικό σημείο, το οποίο αφορά την Ιερουσαλήμ και την απόπειρα που γίνεται να παρεμποδίζετε τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν. Δεν μπορούν να πάνε εκεί που θέλουν. Αποπειράστε να κατεδαφίσετε το τζαμί Αλαξά. Ο πρέσβης μίλησε για την ασφάλεια του Ισραήλ. Γιατί δεν μιλάτε όμως και για τα μέτρα ασφαλείας τα, τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν για να προστατευθούν οι Παλαιστίνοι. Γιατί ταπεινώνονται στα φυλάκια και στα σημεία περάσματος κάθε μέρα. Γιατί ο στατός του Ισραήλ δολοφονεί Παλαιστίνιους στα σπίτια τους και στα εδάφη τους. Γιατί δεν μιλάτε για μέτρα ασφαλεία για του Παλαιστίνιου πολίτε. Επίση, μιλήσατε για την τρομοκρατία. Ομολογώ ότι υπάρχει τρομοκρατία. Σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανώσεων. Αλλά ξεχνάτε την κρατική τρομοκρατία, κύριε Πρέσβη, που είναι η χειρότερη μορφή τρομοκρατία. Μιλάμε για την ε, κατοχή. Η κατοχή είναι τρομοκρατική δράση. Γιατί δεν μπαίνετε σε λεπτομέρειες. Γιατί δεν μιλάτε για τα βασικά σημεία που είναι η ρίζα του κακού. Τα βασικά αυτά σημεία είναι η κατοχή, η κατοχή, η κατοχή. Θα είμαι σύντομος. Σας παρακαλώ δώστε μου ακόμα ένα-δύο λεπτά. Σας παρακαλώ να κλείσετε, να καταλήξετε. Ναι, βεβαίως. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε η Αμερικανή εκπρόσωπος, την ε, ευχαριστώ για όσα είπε. πιστεύουμε ότι πραγματικά υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική της νέας κυβέρνησης. Αλλά πιστεύουμε ότι η αρχική αυτή ορμή ε, κάπως έχει μειωθεί όταν η Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για επικισμούς. Είναι δυνατόν να γίνουν διαπραγματεύσεις ε, αν συνεχίζονται οι επικισμοί. Στην αρχή είχαν πει οι Αμερικανοί ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι κάπως το πήραν πίσω. Νομίζω ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν ε, κράτησε την στεναρή στάση. Επίσης το 1967 οι Αμερικανοί είχαν καταδικάσει την ε, Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινίων εδαφών. Νομίζω ότι σε κάποια φάση είχαν πει ότι πρόκειται για εδάφη όπου υπάρχουν συγκρούσεις. Ε, το ίδιο και με την Ιερουσαλήμ. Είναι ένα χώρο όπου, όπου υπάρχουν συγκρούσει. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί λένε και ξελένε. Θα ήθελα να λένε κάτι και να δεσμεύονται με αυτό. Σε ό,τι αφορά του Ευρωπαίου φίλου, καταλαβαίνετε την κατάστασή μα, το ξέρω, αλλά μερικέ φορέ οι δικέ σα θέσει ε, απηχούν τι απόψει των Αμερικανών. Ελπίζω ότι ο ρόλο σα θα είναι πιο θετικό εφ' εξής σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής και θα βοηθήσετε πραγματικά για να επιληθεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Επίσης, διαβάσαμε και μελετήσαμε την έκθεση Goldstone. Δεν ήταν τόσο θετική. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αν όλοι έκαναν το ίδιο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να οργανώσουμε τη συζήτησή μας. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Φλότρο. Θα ακούσουμε ακόμα μερικές παρεμβάσεις και μετά οι συγκητές μας θα μπορέσουν να απαντήσουν. Ελέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο. Είναι αλήθεια, όπως πάρα πολύ καλά το είπε η θα ξαναπούμε μεταξύ μας αυτά που έχουμε ήδη πει και ξαναπεί τόσες και τόσες φορές μέχρι τώρα. Όμως παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ναι, κάποια νέα στοιχεία. Και αυτό μετά, όχι από έναν πόλεμο, αλλά από μια θανατηφόρα επίθεση των Ισραηλινών στη Γάζα. Αυτό που για μένα είναι προφανέ είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πολλέ συζητήσει, διπλωματικά, πολιτικά, να λέμε ένα σωρό πράγματα για το μέλλον τη Μέσης ανατολή του κόσμου. Υπάρχει όμω κάτι στοιχειώδε. ότι υπάρχουν κάποιε προδιαγραφέ διεθνεί, υπάρχει ένα δίκαιο, διεθνέ δίκαιο. Όταν αυτά παραβιάζονται πρέπει κανεί να βγάζει συμπεράσματα και πρέπει να φροντίζει η κατάσταση πλήρου ατιμορρησία που υπάρχει εδώ και τόσα πολλά χρόνια στην περιοχή να πάψει. Η έκθεση Goldstone αυτό βέβαια είναι για τον κύριο Ρίτμπεργκ να μα πει. Δεν ξέρω αν κατάλαβα πολύ καλά αυτά που είπατε, αλλά εσεί τι θέλετε να πείτε. Για την έκθεση μιλάτε για τον εισηγητή. Τι. Εδώ υπάρχει μια έρευνα συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη, με επιχειρήματα, που στο κάτω-κάτω βάζει και τι δύο πλευρέ. Ε, γιατί και οι δύο πλευρέ αμφισβητούν τελικά την έκθεση αυτή, που είναι καλό σημάδι μάλλον. Λοιπόν όλα αυτά για το ότι η Ένωση, τα κράτη της Ένωσης θέλουν, δεν θέλουν την έκθεση αυτή ανθρώπινα δικαιώματα στη Γενέβη, ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω, έχω ή μάλλον υπερβολικά καλά καταλαβαίνω. Τελικά, δεν πρέπει να έχουμε κάτι χρήσιμο για να προχωρήσουμε, δεν πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα, να πούμε ότι η ατιμορρησία σταματάει, δεν έχει μέλλον όταν πρόκειται για ε, συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ αυτό περιμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό περιμένω από τι Ηνωμένε Πολιτείες, αυτό να πούν και να φροντίσουν να βγουν τα συμπεράσματα που πρέπει. Φοβάμαι όμω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά, γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχει μια συνενοχή εδώ. Έπειτα μπορούμε εύκολα να βγάζουμε ρητορικού λόγου υπέρ τη Ειρηνή, όμω κάποια στιγμή πρέπει να αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα. Δεύτερον, Εκνευρίζομαι πάντα και στο κάτω-κάτω φαίνεται από τον τρόπο που μιλάω. Ε. Εκνευρίζομαι λοιπόν όταν ακούω τον πρέσβη του Ισραήλ να μας μιλάει για τη λωρίδα της Γάζας και να μας λέει αποσυρθήκαμε από την λωρίδα της Γάζας. Ναι, αποσυρθήκατε για να μην κλειστείτε σε αυτή την φυλακή που είναι η Γάζα. Ε. Λοιπόν, μας λέτε φύγαμε από τη λωρίδα τη Γάζας. Μα όχι, όταν κάποιο αποσύρεται, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αφήνει αυτούς που ζουν εκεί ελεύθερα να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει αποσύρωμαι, δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Συνεπώ. πρέσβη Κυριέλ, αναλάβετε τις ευθύνε σα. Μη λέτε ότι αποσυρθήκατε από τη λωρίδα της Γάζας, αφού την κλείσατε. Έπειτα, δεν θα έπρεπε κανείς να κάτσει να σκεφτεί. Ε, λέμε οδικοί χάρτες, δεσμεύσεις που δεν τηρούνται. Ναι, α μετά από όλα αυτά, τι. Υπάρχει το Παλαιστινιακό κράτος. Μήπως πρέπει να τα κάνουμε ανάποδα. Ρωτάω τους εισηγητές. Μήπως θα έπρεπε η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πρώτα να δηλώσει τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους και μετά να ξεκινήσουν να συζητάμε για τους επικισμούς, τα Ιερουσόλυμα κλπ. κλπ. Μήπως θα ήταν αυτή μια μέθοδος πιο καλή που θα δώσει περισσότερα αποτελέσματα. Γιατί στο κάτω-κάτω μέχρι τώρα τι κάνουμε. Γερνάμε και δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Εγώ θα ήθελα να δω ένα Παλαιστινιακό κράτο και ένα κράτο του Ισραήλ να ζουν ειρηνικά δίπλα το ένα στον άλλον. Μήπω λοιπόν να ανατρέψουμε τι προτεραιότητε. Ευχαριστώ κύριε Φλότρο. Όντω ήσασταν πολύ σύντομοι. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ελχαλιφά από την Ιορδανική Αντιπροσωπεία. Και επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω να είσαστε σύντομη και συνεκτική. Μετά η κυρία Νταγκή από την τουρκική αντιπροσωπεία και μετά θα δώσω το λόγο στους εισηγητές για να απαντήσουν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου ευθύ εξ αρχής να εκφράσω τα αισθήματα πελπισίας που νιώθουμε στην περιοχή εξαιτίας ε, της ε, διακοπής της ειρηνευτικής διαδικασίας που κανονικά έχει ξεκινήσει από τη Μαδρίτη. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στην έλλειψη δράσης από πλευράς του Ισραήλ προκειμένου να φτάσουμε σε μια συνολική λύση. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει στο Ισραήλ να ασκεί βία κατά των Παλαιστινίων. Δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχει τέτοια κατοχή, δεν έχει δικαίωμα το Ισραήλ να ασκεί βία. Παρά την κατοχή. Και δεν πρόκειται μόνο για κατοχή, πρόκειται για μια αλλαγή ταυτότητας, πρόκειται για μια αλλαγή στη γη, μια προσπάθεια να γίνει εβραϊκή η γη αυτή. Οι διάφοροι αποσχιστικοί πόλεμοι από πλευράς των ακραίων έχουν χτιστεί ακριβώς πάνω σε αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε απελπισία και σε ακραίες θέσεις. Αυτά ζει ο κόσμος επιτόπου που θέλει μια αξιοπρεπή ζωή. Ο στόχος για τους Ισραηλινούς είναι απλά διαπραγματεύσεις, όχι όμως ειρήνη. Δεκαετίες πέρασαν και ακόμα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της ειρήνης, παρά τις επανελειμμένες διαπραγματεύσεις. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα από τα τελευταία γεγονότα στη Γάζα, για παράδειγμα, ότι η ειρηνική συνύπαρξη είναι ένα στόχος στον οποίο πιστεύουμε εμείς στην Ιορδανία. Αυτός είναι ο στόχος για τον οποίο δουλεύουμε εμείς. Αυτό θέλουμε. Και όχι μόνο να μιλάμε για συνολική ειρήνη, θέλουμε δικαιώματα στην αξιοπρέπεια για όλους. Αλλιώς η κατοχή είναι ο δρόμος για όλα τα δεινά. Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε πλήρης διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προκαθορισμένα πράγματα. Πάυση των επικισμών συμφωνούμε με την αμερικανική άποψη. Έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Συμφωνούμε και με την Ευρώπη επίσης. Και με την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Δαγκέπτου και κυρία Καλημέρα σας και ευχαριστώ. Και καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις ελπίδες ε, που τρέφω για την ε, πορεία προς την ειρήνη. Ότι αυτή δηλαδή η συνάντηση θα μπορέσει να συμβάλλει αποφασιστικά στην ειρήνη. Είμαι πολύ ικανοποιημένη για, τα, για τις εξελίξεις που ακούω και τον Ιούνιο από ό,τι φαίνεται η Αίγυπτος ε, ε, μαζί με την ε, ε, η Ορδανία θα μπορέσουν να οργανώσουν συζήτηση για τα θέματα της Γάζας. Είχα προτείνει λοιπόν να επισκεφθούμε την περιοχή, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Είχαμε προτείνει να γίνει μια fact-finding mission. Πήγα στην περιοχή και βλέπω ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη επίσκεψη και στη Ράφαλα και στην ε, Ιερουσαλήμ όπου είδαμε κυρίως για τη Γάζα με χωρίς κανένα συγκάλυμα την εικόνα της καταστροφής. Ιδιαίτερα οι, εργάτε, οι εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών, οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών στην ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή της ε, Γάζας, οι εκπρόσωποι ε, του Νομοθετικού Συμβουλίου αναφερόμενοι στις τους βομβαρδισμούς του Ιανουαρίου ε, μας έδειξαν ε, πόσο μεγάλες καταστροφές προκάλεσαν αυτοί οι βομβαρδισμοί. Φεύγοντας από την περιοχή είχα σφιγμένη την καρδιά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε μέσα από συναντήσεις όπως σημερινή να ε, αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Τώρα πια, όπως είπε και ο κύριος Προεδρευτής, δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρηση. Πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δεινά. Και σημειώνω ότι η Τουρκία είναι ένα πρότυπο που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλα κράτη Εγώ προσωπικώς επιστρέφοντας στην πατρίδα μου ζήτησα ραντεβού και συναντήθηκα με τον πρεσβευτή του Ισραήλ για να συζητήσω μαζί του τα θέματα της Γάζας. Βλέπω λοιπόν, όπω άλλωστε ακούσαμε και από τον Ισραηλινό προσβευτή εδώ, ότι και εκεί ε, και στην Τουρκία ο Ισραηλινός Προσβευτή μίλησε για την υπόθεση τη Λόρδας της Γάδας, σαν να ήταν μόνο ένα ζήτημα τρομοκρατία και καταπολέμηση τρομοκρατία αποκλειστικά, χωρί καμία διάκριση. Ωστόσο έχω να πω ότι με επηρέασαν πολύ οι συνεντεύξεις που άκουσα την εποχή εκείνη, το 2009, από τον ε, πρεσβευτή του Ισραήλ ε, στην Άγκυρα, ο οποίος μάλιστα έχει γεννηθεί τυχαία στην Τουρκία, ο οποίος έχει ε, περάσει τα χρόνια αυτά στην Τουρκία λόγω εξορίας επιβεβλημένης από τις συνθήκες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μας έλεγε λοιπόν, η διάβασα μάλλον στην έντευξή του, ότι είχε πολύ θετικέ αναμνήσεις από την Τουρκία κτλ. Και του είπα του πρεσβευτή αυτού, όταν συναντηθήκαμε, ελπίζω κάποια μέρα τα παιδιά στη Γάζα μεγαλώνοντας να μπορούν να έχουν θετικές αναμνήσεις για, τις, ε, για τα χρόνια που θα έχουν περάσει εκεί. Ότι θα μπορέσουν δηλαδή να λένε και εμείς περάσαμε ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Με συγχωρείτε, λέει η Έχουν δικαίωμα και τα παιδιά αυτά σε μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία και είπα στον πρεσβευτή ε, του Ισραήλ ότι η Τουρκία αντιμετώπισε πάρα πολλές επικρίσεις για την ανθρωπιστική κατάσταση, για τους βασανισμούς ε, και την παράδοση των ανθρωπινών δικαιωμάτων ύστερα από το πραξικόπημα του 2080. Του είπα λοιπόν ότι ναι, εκφράστηκαν επικρίσεις κατά της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή η οποία επικρίθηκε πολύ από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα έχει πάρει τη θέση της μέσα στα δημοκρατικά κράτη. Και ελπίζω μια μέρα και το Ισραήλ να μπορέσει να έχει μια θέση ισότιμη. Εμείς προβάλλουμε πάντοτε τα δικαιώματα των ε, Παλαιστινίων, αλλά πάνω απ' όλα για μένα έχει σημασία το να αναγνωρίσουμε και τα δικαιώματα του Ισραηλινού λαού, γιατί και εκείνος ε, πολλές φορές ε, λησμονείται, πολλές φορές αντιμετωπίζεται ε, μέσα από την ε, παράνοια για ασφάλεια κατά τρόπο καταπιεστικό. Πολλές φορές περιστέλλονται τα δικαιώματά του στο όνομα της αντιμετώπισης τρομοκρατίας. Τόσο λοιπόν για τους Ισραηλινούς, για τον Ισραηλινό λαό, αλλά και για τον Παλαιστινιακό. Ώστε να απαλλαγεί από αυτή την παράνοια της προβολής της ασφάλειας, των όρων ασφάλειας ο Ισραηλινός λαός, ελπίζω να βρεθεί η λύση. Με συγχωρείτε για την συναισθηματική φόρτιση, αλλά βλέποντα ε, μπροστά στα μάτια μου και πάλι τι σκηνέ που αντιμετώπισα στη Γάζα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Τώρα λοιπόν, Θέλω να σημειώσω μια άλλη διάσταση ότι όταν μιλούμε για ασφάλεια, λησμονούμε ότι έχουμε να κάνουμε με την ανθρώπινη ζωή, ότι εδώ πέρα έχουμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων αυτών. Και εμείς όντας μια χώρα που ζει μέσα σε μια περιφέρεια που αγωνίζεται για τη δημοκρατία αλλά και για την ασφάλεια, για την επιβίωση της, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φορές διπλά μέτρα και σταθμά. Για μας θα πρέπει να σταματήσει αυτό και ανα πάσα στιγμή θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Αυτό είναι ο αγώνας μας. Όπως είναι ο αγώνας της Τουρκίας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενδυναμώσει τη δημοκρατία της, να συμβάλλει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Πρέπει η Ευρώπη να προασπίσει τη δημοκρατία στην περιοχή, την ειρήνη στην περιοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρόπο απόλυτα ειλικρινή και σαφή. Γιατί τώρα η αντιπαράθεση είναι δεδομένη το πεδίο της ρήξης και της σύγκρουσης είναι ζωντανό και δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη. Και ελπίζω και ο Πρόεδρος Ομπάμα να συμβάλλει, όπως είχε δηλώσει αποφασιστικά, στην ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. και πιστεύω ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα με βάση την κοινή λογική οι αρχές του Ισραήλ να σταματήσουν να συνδέουν οποιαδήποτε επίκριση εκφράζεται κατά του Ισραήλ με τον αντισημιτισμό και να δεχθούν να εξετάσουν με λογική όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Εμείς, όπως είπα, η Τουρκία έχουμε υποστεί πάρα πολλές επικρίσεις. Τουρκία, στο Ισραήλ Τώρα βλέπουμε ότι εκφράζονται πολλές επικρίσεις και θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι ώστε να αναπτυχθεί η περιοχή κατά τρόπο ειρηνικό και δημοκρατικό. Ευχαριστώ κύριε Ταγκή. Θα δώσω το λόγο στον πρέσβη, τον κύριο Κουριέλ, εν συνεχεία στον κύριο Ρίτμπεργκ, προς τον οποίο απευθύνθηκαν κάποιες ερωτήσεις και εν συνεχεία στη Λέιλα Σαχίντ. Θα μιλήσω εβραϊκά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα μεγάλη υπομονή και ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός. Όλα όσα ακούστηκαν τα παίρνω πολύ στα σοβαρά. Αλλά θα πρέπει να σας πω επίσης ότι δεν με εκπλήσετε κιόλας. Από την εμπειρία που έχω σε τέτοιου συνεδριάσεις ε, Πραγματικά δεν με εκπλήσουν τα όσα άκουσα. Αλλά παρόλα αυτά ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός. Άκουσα πολλά ερωτήματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Νομίζω ότι είμαι ότι μειοψηφώ αριθμητικά. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να απαντήσω ε, σε όσον τον περισσότερες ερωτήσεις. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά θέματα. Δεν άκουσα τίποτα από τον Αιγύπτιο εκπρόσωπο, τον κύριο Σάσλι, τίποτα το θετικό σε ό,τι αφορά τον ορισμό ε, ή τον προσδιορισμό των δύο κρατών. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε την κατοχή. Ε, αγαπητοί Άραβες, ε, νομίζω ότι η τον προσδιορισμο των δυο κρατων εμεις ειμαστε ετοιμοι να σταματησουμε την κατοχη ε αγαπητοι αραβες νομιζω οτι η απαντηση στα ερωτήματα που σας έχω θέσει δεν είναι σαφής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα συζητάμε τα συμπτώματα αυτού που συνέβησαν, που συνέβησαν μετά τον πόλεμο των ε, έξι μερών, μετά το 1967. Πριν το 1967 δεν υπήρχε κατοχή, δεν υπήρχαν κατεχόμενα εδάφη. Επομένως και δεν υπήρχε και, και ειρήνη. Ένας από τους βασικούς λόγους που συζητιέται και στις διαπραγματεύσεις είναι ότι οι Παλαιστίνοι και οι Άραβες είναι το ερώτημα είναι μάλλον, είναι έτοιμοι να αναγνωρίσετε το Ισραήλ ως εθνικό κράτος του Ισραηλινού λαού. Αν πάρετε την ε, παλαιστινιακή θέση που λέει ναι σε δύο κράτη, ναι στη λύση των δύο κρατών, αλλά παράλληλα θα υπάρξει μια επιστροφή εκατομμυρίων προσφύγων στο Ισραήλ, μιλάμε για Παλαιστίνιους ε, πρόσφυγες. Αυτό στην πραγματικότητα είναι σαν να αρνείστε ουσιαστικά τη λύση των δύο κρατών. Παράλληλα το Ισραήλ δεν ζητάει ε, ως προϋπόθεση την αναγνώριση του Ισραήλ ως εθνικό κράτους ε, του, των Ισραηλινών. Δεν ζητάμε να γίνει προϋπόθεση αυτή για τις διαπραγματεύσεις. Και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Λέιλα Σαχίδ ότι η Γκάζα ε, είναι τμήμα της Παλαιστίνης και πληθυσμιακά αλλά και εδαφικά. στο εσωτερικό των Παλαιστίνιων υπάρχουν τόσες πολλές ε, διαφωνίε. Αν δεν υπάρχει ενότητα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξανά για αυτό το θέμα. Γιατί μπορούμε να με, το... με τη Γάζα δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Αμαχουμταμπάς, με την ε, Δυτική Όχθη, αλλά δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με τη Γάζα. Και παρόλα αυτά δεν τα θέτουμε αυτά ω προπόθεση για τι διαπραγματεύσει. Το είπα αυτό στην παρουσίασή μου. σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται ε, να τονιστούν ας πούμε, οι αδυναμίες των άλλων. Εγώ δεν μπαίνω. Δεν θέλω να, να υπογραμμίσω τις αδυναμίες των Παλαιστινίων. Υπάρχουν αδυναμίες που θέτουν ε, ερωτηματικά ε, για την επίτευξη μια συμφωνίας. Αν όχι τόσο για την επίτευξη, τουλάχιστον για την ε, πρακτική υλοποίηση των διατάξεων αυτής της συμφωνίας. αν ένας ε, εξωγήινο έφτανε στην αίθουσα εδώ <laughs> σήμερα το πρωί, θα, πίστευε ότι τα προβλήματα είναι μονόπαντα, από τη μία πλευρά μόνο. Εμείς, και, και εμείς οι Ισραηλοί, είμαστε απογοητευμένοι από το γεγονό ότι μέχρι τούδε διαπραγματεύσεις δεν έφεραν καρπού. Θέλαμε και εμείς την ειρήνη. Σήμερα ακούω τον πρόεδρο Μαχμούτα Μπάς να λέει ότι λυπάται για το γεγονός ότι δεν δέχτηκε τις προτάσεις του Προέδρου του Πρωθυπουργού, συγγνώμη, Όλμερτ. Ε, πρέπει να γνωρίσουμε όλοι μας ε, τα λάθη μας, το, να κάνουμε όλοι μας ε, το μια κούλπα. Εμείς, θέλω να, επανέλθω στη Γάζα, φύγαμε από την Γάζα. Θέλουμε η Γάζα να γίνει ένα θετικό μοντέλο που θα έχει επιπτώσει σε, όλες τις, ε, σε όλο το φάσμα των διαπραγματεύσεων. Φύγαμε από τη Γάζα και θέλουμε οι Παλαιστίνοι να διαχειριστούν την ύπαρξή τους στη Γάζα χωρίς κατοχή. Επανέρχομαι στο παράδειγμα που έχω ξαναδώσει πολλές φορές στη Γάζα ε, δώσαμε, αφήσαμε, κληροδοτήσαμε ε, θερμοκήπια. Ε, σας δώσαμε τη δυνατότητα να καλλιεργήσετε ε, φρούτα και λουλούδια και να τα, να τα εξάγετε ε, προς την Ευρώπη. Υπάρχουν αυτά τα θερμοκήπια, θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν οι Παλαιστίνοι, θα μπορούσαν να βρουν δουλειά ναι, θα μπορούσαν να εργαστούν σε αυτά τα θερμοκήπια. Δύο εβδομάδες μετά από την απόσυρση των Ισραηλινών από τη Γάζα δεν υπήρχε ούτε ένα θερμοκήπιο. Καταστρέφηκαν. Μπορούμε να, κατηγορούμε τους άλλους, το Ισραήλ, ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που κάνατε. Κάποια πράγματα που οι Παλαιστίνοι θα μπορούσαν να κάνουν για τον εαυτό τους, για το καλό τους. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση στη Γάζα ή το, το φράγμα αυτό της ασφάλειας που αναφέρεται. Είπαμε, είπατε μάλλον ότι ξαφνικά το Ισραήλ ας πούμε ξύπνησε και είπε «Α, τι θα κάνω μια επιχείρηση στη Γάζα». Κύριε Βέγγελ, συμφωνώ ότι ίσως δεν σας ξεκαθάρισα κάποια πράγματα καλά. Ίσως δεν εκφράστηκα καλά. Ε, σε καμία περίπτωση ε, όλοι οι κάτοικοι της Γάζας, όλα τα παιδιά και οι γυναίκες είναι αλλά είναι σαφές, είναι γεγονός ότι ελέγχεται η Γάζα από μια τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό ήθελα να πω. Είναι υπό τον έλεγχο μια τρομοκρατική οργάνωση. Γιατί η Χαμά είναι τρομοκρατική οργάνωση και υπάρχει και στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Αυτό είναι σημαντικό. Η Χαμά χρησιμοποιεί τρομοκρατικέ ε, δράσει και εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Επί, επί 8 χρόνια βομβάρδισε με πυράβλους με όλμους δεκάδες ε, Ισραηλινά χωριά γύρω από τα σύνορα. Ε, το να λέτε ότι ένα πρωί ξυπνήσαμε και αποφασίσαμε να εισβάλλουμε στη Γάζα νομίζω ότι είναι διαστρέβλωση της αλήθειας. Ε, δείξαμε φοβερή ε, υπομονή επί 8 χρόνια ε, για τη Γάζα. Ε, δεν είχαμε άλλη επιλογή, έπρεπε να υποστηρίξουμε και να υπερασπιστούμε τους αμάχους. Λυπόμαστε για τους θανάτους στη Γάζα, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο σαβαρά. δεν είναι τόσο απλά. Επίση, αυτό το, το φράγμα τη ασφάλεια δεν δημιουργήθηκε έτσι μία νυχτή. Μετά από χρόνια ε, επιχειρήσεων των ε, καμικάζι αυτοκτονία ε, στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, στην, στη Ράφα, σε διάφορες περιοχές χρειάστηκε να υψώσουμε ένα φράγμα μεταξύ των οχημάτων που ερχόταν από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, τα οποία ανατινάσσονταν στο εδάφό μας. Δεν είναι κακή πίστη αυτή απέναντι στο, στους Παλαιστίνιους από πλευράς μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι των αντεγκλήσεων, των αμοιβαίων αντεγκλήσεων, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά αρνητικό. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει θετική και ενδιαφέρουσα αν κοιτούσαμε προ τα εμπρό, το μέλλον, αν αποφασίζαμε ότι είναι σημαντικό το να διαπραγματευτούμε, το να αναγνωρίσουμε την ιστορία, να αναγνωρίσουμε την επίσημη ιστορία της άλλης πλευράς, να αναγνωρίσουμε ότι καμία πλευρά δεν έχει απόλυτα δίκιο ή απόλυτα άδικο. Μπορούμε να μιλήσουμε για το νερό, μπορούμε να μιλήσουμε και για την Ιερουσαλήμ. Μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες ε, δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην Ιερουσαλήμ. Ε, ποτέ δεν υπήρχε ε, από το 67 και μετά τέτοια θρησκευτική ελευθερία όπως σήμερα. Υπάρχουν προκλήσεις στην Ιερουσαλήμ από την αραβική πλευρά που αποφάσισε να παροτρύνει τους ε, πιστούς μουσουλμάνους ε, προς τη βία. Νομίζω ότι το Ισραήλ έχει την πρόθεση να διατηρήσει τη θρησκευτική ελευθερία όλων των κοινοτήτων. Όπω το έκανε από το 67 και μετά. Δεν έχει κανένα ε, συμφέρον το Ισραήλ να υπάρχουν εξεγέρσεις στην Ιερουσαλήμ σε καμία περίπτωση δεν είναι προ το συμφέρον μα. Δεν ξέρω να απάντησα σε όλε τι ερωτήσει, γιατί ήταν πάρα πολλέ. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να φύγουμε από εδώ με έτσι μια πιο αισιόδοξη διάθεση. Νομίζω ότι ο Παλαιστίνιος λαός έχει εξαιρετικές ικανότητες και νομίζω ότι το Ισραήλ επίσης έχει εξαιρετικές ικανότητες. Πιστεύω ότι κανένας από τους εταίρους δεν θα κερδίσει από την ε, διαιώνιση της ε, ε, του πολέμου. Γιατί μα το λένε οι άλλοι, αλλά γιατί είναι για το συμφέρον και το δικό σα, αλλά και κυρίω το δικό μα, να σταματήσει αυτή η σύγκρουση, να υπάρξουν δύο κράτη δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι δύο λαοί, ο Παλαιστινιακό λαό και ο Ισραηλινό λαό, μπορούν να βελτιώσουν την ύπαρξή του πολύ περισσότερο από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ε, η εκπρόσωπος της Τουρκίας τα είπε πολύ σωστά αυτά τα πράγματα. Το παράδειγμα της Τουρκίας θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε τα προβλήματα ε, για το νερό μεταξύ Ισραήλ και Αράβων. Αν δούμε το υδάτινο δυναμικό, το ειρηνευτικό δυναμικό που υπάρχει, το τουριστικό δυναμικό, πραγματικά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ε, νομίζω ότι οι διαπραγματεύσει από το και μετά δεν ήταν απώλεια χρόνου. Νομίζω ότι σήμερα έχουν καταλάβει όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι Όλοι μιλάμε για το ίδιο πράγμα τελικά. Θα πρέπει τα δύο μέρη να εφαρμόσουν από κοινού αυτή τη λύση. Και πιστεύω τότε, όταν υπάρξει αυτή η κοινή λύση, θα υλοποιηθεί και αυτό το θετικό δυναμικό. Αν ξέχασα κάποια ερώτηση, παρακαλώ υπενθυμίστε μου τι. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρέσβη, θα ξαναπάρετε το λόγο αργότερα. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Σέιντ, η οποία πρέπει να φύγει σε πέντε λεπτά. Και μετά ο κύριος Ρίτμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, δυστυχώ, πρέπει να φύγω σε λίγο. Γι' αυτό και παίρνω το λόγο πριν από τον πρέσβη Ρίτμπεργκ. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι εδώ υπεύθυνοι άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα. Θα ήταν έλλειψη σεβασμού απέναντι στους εκλεγμένους βουλευτές να ξεχνάμε ότι έχουν αρκετές πληροφορίες για να γνωρίζουν, κύριε Κυριέλ, την πραγματικότητα. Τώρα αν εσείς έχετε την αίσθηση για κάτι διαφορετικό, Ίσως είναι γιατί έρχεστε από την μόνη χώρα που στον 21ο αιώνα κατέχει μια άλλη χώρα. Και αυτό εδώ και 40 χρόνια και με παραβίαση όλων των κανόνων δικαίου. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνετε ότι το καταλαβαίνει και είναι κάτι προφανές για οποιοδήποτε κοιτάζει σήμερα την τηλεόραση, διαβάζει εφημερίδες, διαδίκτυο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Εγώ να δεχτώ την πραγματική σας θέληση για ειρήνη στην Ισραηλινή κοινωνία. Πραγματικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει την ειρήνη. Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτή και η βούληση της σημερινής Ισραηλινής κυβέρνησης. Γι' αυτό και λέω, ακόμα και αν δεν έγιναν πολλές ερωτήσεις άμεσα για το άτομό μου, εγώ θα πω ότι αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε, που δεν είναι ακόμα πραγματικότητα βέβαια, δεν εξαρτάται μόνο από εμά, εξαρτάται και από τους διεθνείς μας εταίρους. Είμαι σε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη ΠΕΜ, που είναι ένα όργανο το οποίο θέλει την ειρήνη, γιατί όλοι στην ΠΕΜ αυτό θέλουμε, αλλά σήμερα ξέρω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε που εκπροσωπεί η κυρία σήμερα έχουν άμεση ευθύνη για την κατάσταση και έχουν την δυνατότητα να πιέσουν για να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις όπως έχει εξηγήσει και ο Πρόεδρός μου σε σταθερές βάσεις με σημεία αναφοράς. Δεν είμαστε έτοιμοι να πηγαίνουμε να διαπραγματευόμαστε σε ένα γενικό φλού, σε οριστίες. Όχι, πρέπει να υπάρχουν να σταματήσουν μάλλον οι προϋποθέσεις της κατοχής, ο επικισμός κύριε Πρέσβη, τι κάνει, δεν μειώνει την κατοχή, την αυξάνει. Οπότε σήμερα, και πραγματικά χαίρομαι που έχουμε, όπως είπε και η Πρόεδρος, ότι πρόκειται για επίσημη ανταλλαγή, αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο, στην Ουάσιγκτον, σε πιο επίσημο επίπεδο από αυτό που είμαστε εμείς εδώ σήμερα, Ελπίζω να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Όλες οι πλευρέ που έχουμε υπογραμμίσει δεν είναι θέμα δικιά μα αντίληψη των Αράβων ή των Ισραηλινών. Το λέει το διεθνές δίκαιο. Αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, εσείς οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, αν εσείς θέλετε να βασιστείτε στο διεθνές ε, δίκαιο, έχει καλώς αλλιώς, είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Και αυτό είναι και το κλειδί για τη βία σε ολόκληρη την περιοχή. Πιστεύω λοιπόν πως σήμερα υπάρχει μια δυνατότητα. Πρέπει όμως να είναι ξεκάθαρη και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του προς τη σωστή κατεύθυνση. Συγγνώμη ζητάω από τους υπόλοιπου, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγω. Euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαΐτ. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Ρίτσπερκ, στον οποίο απευθύνθηκε η κυρία Φλότρο. Και πρέπει να σας πω ότι έχω κατακλειστεί από σημειώματα, όπως αυτό. Όλοι θα λάβουν το λόγο. Αλλά ο κύριος Ρίτπερκ πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στην έκθεση Goldstone, που όπως όλοι γνωρίζουμε έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Η έκθεση προκύπτει ύστερα από έναν τραγικό πόλεμο. Ο πόλεμος είναι πάντα τραγικός, αλλά αυτό ήταν άκρος τραγικός, τόσο πολιτικά όσο και ανθρωπιστικά τραγικός. Η απόφαση για τη σύνταξη της έκθεσης ελήφθη από ένα σώμα το οποίο έχει παρελθόν μακρό. Εδώ θα εντολή κατά την άποψη Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι ισορροπημένη διότι επικεντρωνόταν μόνο στο ένα μέρος της ε, σύγκρουσης. Πλην όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε και την ε, ικανοποίησή της ως προς την επιλογή του Προέδρου της Επιτροπής, γνωστού, ανεγνωρισμένου και ανεξάρτητου δικηγόρου. Είδαμε επίση με ικανοποίηση την απόφαση του ίδιου του Προέδρου ε, που έκρινε ότι είναι σκόπιμο να επεκταθεί η εντολή ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές της σύγκρουσης για την άποψή μα ήταν σφάλμα τη Ισραηλινής κυβέρνηση το ότι απέριψε την πρόταση για συνεργασία με την Επιτροπή αυτή εκ, των, εκ προημίου. Συνέπειες αυτής της επιλογής είναι όλα αυτά τα οποία είδαμε έκτοτε. Η έκθεση πραγματεύεται πολύ σοβαρά ζητήματα, κατά τρόπο πολύ σοβαρό, και εκφράζοντας πολύ σοβαρές κατηγορίες και με σοβαρότητα. Η συζήτηση που ανέπτυξαν τα ευρωπαϊκά κράτη ως προς την έκθεση αυτή, περί την έκθεση αυτή είναι και όπως γνωρίζετε ασφαλώς γιατί παρακολουθείτε και τις συζητήσεις στις διάφορες χώρες κάπως διαφορετική. Ανακράτος μέλος δηλαδή υπάρχουν διαφορές, γνωστό αυτό, καθήκον της Προεδρίας ήταν να προσδιορίσει μια κοινή ευρωπαϊκή θέση και πιστεύω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι παρά τις ε, μάλλον δύσκολες εσωτερικές συζητήσεις ε, μπορέσει να βρούμε συνένεση σε διάφορα ουσιώδη ζητήματα τα οποία, στη, τη συνένεση την οποία έχουμε ε, μεταφέρει στις συζητήσεις μας στη Γενέβη και θα συνεχίσουμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Είμαστε ενωμένοι και απερίφραστα δηλώνουμε ότι δεν επιτρέπεται ατιμορρησία σε περίπτωση παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Κάθε τέτοιου είδους ισχυρισμός θα πρέπει να διερευνάται διεξοδικά και στη Γενέβη όπως άλλωστε και στη Νέα Υόρκη, υπογραμμίσαμε με έμφαση ότι την πρώτα αρχική ευθύνη για τη διερεύνηση των παραβιάσεων αυτών τη φέρουν τα ίδια τα μέρη. Πρόκειται για μια βασική αρχή του διεθνούς δικαίου. Θέλουμε, αναμένουμε την συνέχεια στην έκθεση ε, Goldstone που θα δοθεί από το ε, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, Ζητούμε, ζητήσαμε από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να ε, μιλήσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ως προς τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στο θέμα αυτό και αντίθετα με τα όσα μερικές φορές αναφέρονται από τον τύπο δεν συμφωνήσαμε δεν συμφωνήσαμε να αποκλείσουμε περαιτέρω μελέτη της εκθέσεως από κάποιο άλλο όργανο και παραμένουμε ενωμένοι στο θέμα αυτό, το βασικό θέμα που είναι συνδεδεμένο με την έκθεση Goldstone, ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας πιστεύω, ότι δηλαδή ο συνεχιζόμενος αποκλισμός της Λωρίδας της Γάζας είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος για λόγους ανθρωπιστικούς, είναι απαράδεκτος για λόγους πολιτικούς και μπορώ να προσθέσω είναι απαράδεκτος για λόγους ηθικούς. Αυτή είναι η στάση μας, αυτή είναι η θέση μας. Αυτό είναι το μήνυμα που θα συνεχίσουμε να μεταδίδουμε στις συζητήσεις μας και, να μεταφέρουμε και, στη, και θα μεταφέρουμε και στη Νέα Υόρκη και τη Γενέβη. Συζητούμε σε στενό διάλογο με τους Παλαιστινίους φίλους και με άλλους και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ κύριε Ρίτπερκ. Ο πρέσβη Κυριέλ θα πρέπει να φύγει και 12.30. Έχουμε ήδη μεγάλη καθυστέρηση σημειώσει. Θα μου επιτρέψετε να λάβω εγώ το λόγο. Θα μου επιτρέψετε. Ευχαριστώ. Θα οργανώσουμε λοιπόν τις συζητήσεις μας κατά τον εξή τρόπο. Δίνω το λόγο κατά προτεραιότητα στις αντιπροσωπείες που δεν έχουν μιλήσει. Εσείς κύριε Μπαζά μπορείτε να λάβετε ένα λεπτό ως δικαίωμα να απαντήσετε στο ζήτημα της ε, αναγνώρισης του Ισραήλ. Οι λοιπές αντιπροσωπείες όμως είναι Μπρέσκη από την Αλγερία, τα Ταμπάρκη από την Τινησία, Αντάτο, Συρία, Πεγιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βέλα από την Μάλτα και ο κύριος Χατζηνικόλας από την Κύπρο και μετά οι άλλες αντιπροσωπείες, μάλλον άλλα μέλη αντιπροσωπιών που έχουν ήδη τοποθετηθεί Κύριε Αμπάζα. Θα ήθελα μόνο να απαντήσω πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε, στα όσα είπε ο πρέσβης Κυριέλ ως προς την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ και τη θέση της Αιγύπτου. Η Αιγύπτος έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ και έχει αναπτύξει διπλωματικές σχέσεις όπως με κάθε κράτος που έχει διπλωματικές σχέσεις στο Ισραήλ ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για την αναγνώριση ενός κράτους. Δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από οποιοδήποτε κράτος να αναγνωρίσει κράτος λευκό, μαύρο, σοσιαλιστικό είμαι. Η αναγνώριση ενό κράτου προβλέπεται με βάση τις αρχέ του δημοσίου διεθνούς δικαίου, με βάση κανόνε και είναι πάρα πολύ σοβαρό το να προσπαθεί κανεί να ξαναανοίξει το ζήτημα τη αναγνώριση Οι πρόσφυγε. είναι ένα ζήτημα που ε, αφορά το κράτος του Ισραήλ, ναι, τα άλλα κράτη, ναι, τα γειτονικά κράτη, ναι, αλλά ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο. Το δημόσιο διεθνές δίκαιο προσφέρει τους απαραίτητους όρους αναφοράς. Η αναγνώριση όμως κράτους με χαρακτήρα άλλων από αυτών των οποίων όλοι έχουν μέχρι τώρα αναγνωρίσει είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Κανένα κράτος στον κόσμο δεν αναγνωρίζει όρος, ε, κράτος υπό ιδιάζοντες όρους. Ούτε είναι δυνατόν να το πράξει αυτό. Ευχαριστώ και το λόγο θα λάβει τώρα ο κύριος ε, Ρέζγι. Παρακαλώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω πολύ σύντομα για το θέμα μας. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις παρεμβάσεις των διαφορών ομιλητών. Θα ήθελα να κάνω μία, μία ερώτηση προς τον κύριο Ριντμπερκ για την έκθεση Coldstone. Ε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι χάνουμε χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που υπόθηκαν και ξαναυπόθηκαν. Και όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και καιρό. Και αν θέλουμε να προχωρήσουμε προς την ειρήνη, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Με τις επιθέσεις εναντίον του λαού της Γάζας, ακούσαμε να χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οντότητα, παρότι ο πρέσβης του Ισραήλ κάπως διόρθωσε την, το χαρακτηρισμό του. Επίσης, ε, μαθαίνουμε για τις επιθέσεις ε, προς ε, θρησκευτικά τεμένη, το Τζαμί Αλαξά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο ειλικρινή και τίμιο. Όταν κάποιος αισθάνεται ότι βιάζεται η αξιοπρέπειά του, αντιδράει όπως να είναι. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας δεν είναι εδώ ε, γιατί του αρνήθηκαν την θεώρηση του διαβατηρίου. Το είπατε εσείς κυρία Πρόεδρε. Ποια είναι τα σημάδια, χειρονομίες καλής θέλησης που θα μας οδηγήσουν προς μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και μια ειρήνη. Η κυρία Λέιλα Σαΐτ μας μίλησε για τους επικισμούς. Ε, κάνουμε κάτι και λέμε το αντίθετο. Μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για διάλογο, για επανέναρξη του διαλόγου και παράλληλα επεκτείνουμε τους επικισμούς παντού στην Παλαιστίνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε τίμοι και σαφείς. Νομίζω ότι αν αυτή η κοινοβουλευτική συνέλευση και η πολιτική επιτροπή θέλει να προχωρήσει, θα πρέπει να υποφεληθούμε από την έλευση στην εξουσία του Πρόεδρου Ομπάμα. Ακούσαμε την Υφυπουργό, την κυρία Κέρτιν, που μίλησε για τις ελπίδες των Αμερικανών. Ας υποφεληθούμε επίσης ε, από τον κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσουμε. Και ας υπάρξει μια πρωτοβουλία αραβική για την ειρήνη. Ε, ας προχωρήσουμε ε, με τις προσπάθειες του, της τετραμερούς. Ας προωθήσουμε τις ε, πρωτοβουλίες του οδικού χάρτη. Ε, είναι σωστό αυτό που, είπε η κυρία Φλότ. Ένας ολόκληρος λαός τιμωρείται και υποφέρει. Δεν θα πρέπει να βομβαρδίσουμε ένα λαό. Ε, δεν είναι σωστό αυτό και νομίζω ότι από αυτού η έκθεση ε, Goldstone ήταν πολύ σαφής. Ο κύριος Ταμπάκη από την Τινησία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν. Ε, ευχαριστώ και συγχαίρω όλους τους συναδέλφους που ήρθαν ε, σε αυτή την Επιτροπή μετά τις τελευταίες εκλογές, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να τονίσω και να συγχαρώ τους Αμερικανούς ε, για τις θετικές προσπάθειές τους για να συνεχιστεί η διαδικασία, για να προχωρήσει η διαδικασία μέσω των ε, διπλωματικών τους δράσεων. Μας βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά την 64η ε, σύνοδο της συνέλευσης του ΟΗΕ, θα ήθελα να πω ότι Αυτή η επιλογή του Προέδρου Ομπάμα να δουλέψει διμερώς με κάθε ένα από τους ενδιαφερόμενους στην ειρηνευτική διαδικασία, νομίζω ότι εγείρει τα ίδια, ε, τα... Τα ίδια, προσκόμα... τα ίδια προσκόμματα. Δεν είναι εύκολο να πετύχουμε έτσι την ειρήνη στην Ιερουσαλήμ και στους επικισμούς. Υπήρχε μια προϋπόθεση για το πάγωμα της επέκτασης των επικισμών και θα πρέπει η ασφάλεια των Ισραηλινών να συνοδευτεί από την απόρριψη της βίας και από την εξομάλυση των σχέσεων Ισραήλ και αραβικών χωρών. Υπάρχει μια αποτυχία της συνόδου της Τριμερούς, στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος Ομπάμα, με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, που σκοπό είχε να παγώσουν ε, τους επικισμούς, αλλά αυτή η απόπειρα δεν πέτυχε, αυτή η απόπειρα της τριμερούς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό μίλησε με δρυμή τρόπο για την διεθνή αναγνώριση της ταυτότητας του Ισραήλ. Χωρίς όμως να έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ καμία από τις δεσμεύσεις των διαπραγματεύσεων. Χωρίς να έχει υπάρξει καμία, κανένα αποτέλεσμα. Όλες αυτές οι Όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια είναι συγκυριακά και οι διαπραγματεύσει θα συνεχιστούν. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι επεκτάσεις των επικισμών, βλέπουμε ότι στο, στην, στο τζαμί του Αλαξά δημιουργούνται προβλήματα, βλέπουμε τι κάνουν οι εξτρεμιστές που, μπορούν, που προσπαθούν να φτάσουν στην πλατεία του Τζαμιού Αλαξά, νομίζω ότι όλα αυτά εντείνουν τις εντάσεις μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Και παρά τις προσπάθειες της Αμερικανικής κυβέρνησης που σηματοδοτούν μια αλλαγή στη στρατηγική, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ομπάμα ανακοίνωσε αλλαγή στη στρατηγική της Αμερικανικής πλευράς, ε, δεν αρκούν οι έμεσες συνομιλίες σε αυτή τη φάση. Δεν αρκούν και μπορεί να σταματήσουν και ο Νούπο. Τότε θα έχουμε ένα νέο κύμα βίας σε όλη την περιοχή, αν σταματήσουν έστω και αυτές οι άμεσε συνομιλίες. Πιστεύω ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να εστιάσει σε απλούς στόχους. Παραδείγματο χάρη το να σταματήσει η επέκταση των επικισμών και να βοηθήσει τις αιγυπτιακές προσπάθειες ε, για να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Ε, με το να δώσει ε, διεθνή προστασία για τους Παλαιστίνιους και να, σταματήσει, να βοηθήσει στο να σταματήσει η συλλογική τιμωρία και οι επιθετικές πολιτικές ε, και να σταματήσει βεβαίως η κατοχή στη λογία της Γάζας. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Τετραμερή, για να υιοθετηθεί μια ευρεία προσέγγιση με σκοπό την επίλυση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης. Επίσης θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και με τη Συρία και το Λίβανο παρα, εκ παραλλήλου. Ευχαριστώ κύριο Σαντάτ, Σύρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο μέχρι τώρα πριν από μένα για αυτό το θέμα. Όντω υπήρχε βοκοτάρισμα εδώ πέρα και είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ μετά την επίθεση στη Γάζα. Ε, θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε για την γενοκτονία αυτή που διαπιστώσαμε στην Γάζα. Δεν θέλαμε και ούτε και σήμερα να έρθουμε εξαιτία τη ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην έκθεση Goldstone. Πάντω, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν απάνθρωπε πρακτικέ που σκοτώνουν κόσμο, καταστρέφουν τέτοιες πρακτικές δεν είναι μάλλον αυτές ε, οι πρακτικές οι οποίες καταφέρνουν να απομονώσουν τις ακραίες θέσεις, αντίθετα τις ενισχύουν. Το να σκοτώνονται με αυτόν τον τρόπο γυναίκες, παιδιά, αυτό ενισχύει τις προσπάθειες των ακραίων. Τους βοηθάει. Κάποιος είπε, κυρία Πρόεδρε, ότι η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη ε, δεν είναι η μόνη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η μόνη σύγκρουση διαπιστώνω ότι η σύγκρουση είναι μία και ίδια που έχει ξεκινήσει εδώ και τόσα χρόνια και συνεχίζεται. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα στη Δυτική Όχθη υπάρχουν 500.000 ε, επικιστές ε, από το Ισραήλ. Είναι μια τακτική που έχει οδηγήσει στο 20% της περιοχής της Δυτικής Όχθης να καλύπτεται από επικισμούς. 15% σημερα τη κάποια στιγμή ήταν 20-15%, λένε ότι μπορούμε να έχουμε ένα κράτος εκεί. Μα είναι δυνατόν σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα να μπορεί κανείς να φτιάξει κράτος. Γιατί συνεχίζουμε και μιλάμε για έναν κρατούμενο. Όταν είχαμε 11.000 κρατούμενους στο Ισραήλ γιατί τότε δεν έγινε τίποτα, γιατί τότε δεν βάζαμε το θέμα. Το μισό από το Παλαιστινιακό Συμβούλιο που είχε εκλεγεί βρέθηκε στη φυλακή. Γιατί δεν το είπαμε αυτό. Όχι. Λένε είναι λίγοι. Γιατί. Όχι γιατί είναι η μειοψηφία, αλλά είναι η μειοψηφία η οποία ξέρει την αλήθεια. Εκείνη είναι η μειοψηφία που ξέρει την πραγματικότητα. Εκείνη που επιτίθενται δεν δίνουν τη λύση. Ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στη σύγκρουση αυτή καλύπτεται από μία αλήθεια, που είναι ότι μία πλευρά δεν θέλει την ειρήνη. Εμείς πάντα θέλαμε την ειρήνη. Για μας αυτό είναι μία σταθερά δεν αμφισβητείται με τίποτα. Αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τίποτα από τη γη μας. Ούτε ένα εκατοστό. Οι επιθυμίες του Ισραήλ απορρίπτονται και από εμά και από ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς θέλουμε μία δίκαια και συνολική λύση για τη Μέση Ανατολή. Ιδίω όταν το Ισραήλ λέει ότι συμφωνεί με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Επούντο. Όλος ο κόσμος είναι εναντίον τους. Όλος ο κόσμος ψήφισε τα ψηφίσματα του... Ε, των Ηνωμένων Εθνών, 438 κλπ. Όμως δεν τα εφαρμόζει το Ισραήλ. Αν το Ισραήλ ήθελε ειρήνη με τους Άραβες, τότε θα έπρεπε να κάνει αυτό που πρέπει για να εφαρμόσουν τα ψηφίσματα αυτά. Ή να σταματήσει τους επικισμούς. Δεν μπορούμε να οδηγηθούμε με την πολιτική που έχουν απέναντι στους επικισμούς σε ειρήνη. Αυτά τα λέω. Επαναλαμβάνοντας ότι εδώ πέρα πρόκειται για σύγκρουση Αράβων Ισραήλ. Δεν είναι μόνο η Παλαιστίνη. Μπορεί να έγιναν κάποια βήματα στο παρελθόν, αλλά δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Η ειρήνη δεν έχει επιτευχθεί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για να υπάρχει μια βιώσιμη και πραγματική λύση πρέπει να υπάρχει ειρήνη. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα Τεροσόλμα. Αυτή θα είναι η πρωτεύουσα. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο. Και οι πρόσφυγες βέβαια. Με αυτό να ξεκινήσουμε και μετά να πάμε στα άλλα. Το Ισραήλ πρέπει να εγκαταλείψει τον Κολάν. Πρέπει να αποσυρθεί γιατί τους ενδιαφέρει. Πρέπει να φύγουν από όλα αυτά τα ε, φυλάκια και να ξεχάσουν την επιθυμία τους να παραμείνουν στο Κολάν. Να φύγουν από το Καφασουβά επίση, στα σύνορα με το Λίβανο. Να, κάποιες προϋποθέσεις, αρχές από τις οποίες δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε. Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα πολύ επικίνδυνο θέμα. Επαναλαμβάνω και λέω ότι η ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει. Τα όσα έγιναν πρόσφατα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Η τελευταία επίθεση που έλαβε χώρα λίγες μέρες μόνο μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, όπου ο Ισραηλινός ο Πρωθυπουργός είπε ότι έβαζε τις, τα θεμέλια για την ειρήνη κλπ. Μα πώς όταν υπάρχουν άνθρωποι που ζουν υπό αυτό το καθεστώς της κατοχής αναγκαστικά πρέπει να πολεμήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Το αντίθετο, θέλουμε την ειρήνη. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφερθεί και το Ισραήλ, λέγοντας σε όλους τους στρατιώτους ότι εμείς θα εφαρμόσουμε όσα λέει το ψήφισμα 438 του ΟΗΕ. Ένα λεπτό δώστε μου ακόμα κυρία Πρόεδρε. Εμείς λέμε στην άλλη πλευρά, ένα λεπτό, ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό μόνο. Λέμε λοιπόν ότι η Μέση Ανατολή είναι σαν ένα ηφαίστειο έτοιμο να κραγεί. Όσο υπάρχει κατοχή θα υπάρχει και αντίσταση. Και διαφωνώ με, τον, ε, με την εκπρόσωπο της Παλαιστινικής Αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι δεν είναι τρομοκρατία, είναι αντίσταση. Μα όσο έχουμε κατοχή θα έχουμε αντίσταση. Εύχομαι κάποια στιγμή να έχουμε ειρήνη στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πηγαίνουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητέ. Ο Ισραηλινός πρεσβεύς προσπάθησε ξεκινώντας να δημιουργήσει ένα κλίμα θετικό, μιλώντας για την ειρήνη και πιστεύω βεβαίως και εγώ ότι ο προλαλής από τη Συρία επιθυμεί την ειρήνη. Ε, πρέπει να ομολογήσω πάντως ότι είναι κάπως παράδοξη η συζήτηση σήμερα. Αν θέλουμε να είμαστε και σοβαροί ως προς μας ε, των βουλευτών, και επιτρέψτε μου να είμαι εγώ η φωνή η οποία θα φέρει κάποιες αντιρρήσεις στη συζήτηση αυτή. Είναι λίγο δύσκολο τις συζητήσεις μας να τις πάρουμε στα σοβαρά, ε, ε, με τον ισχυρισμό δηλαδή ότι επιθυμούμε την ε, ειρήνη, ισχυριζόμενοι ότι είναι μια, ένα κράτος καταπιεστικό, ένα κράτος που μόνο κάνει, έχει κατοχή και εισβολή και παραβιάζει κάθε τους ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα εκπλήσουμε πάω τον κύριο Ελσαΐτ, παλιό φίλο από χρόνια, ο οποίος είπε ότι είναι εις βάρος της επιβίωσης του Ισραήλ η παρουσία του. Νομίζω ότι πολλά κράτη θα μπορούσαν να διδαχθούν αντιθέτως από τα δημοκρατικά, για τα δημοκρατικά δικαιώματα από την ε, πορεία του Ισραήλ μέχρι τώρα. Επίσης θέλω να πω ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί οι εγγύησεις για την επιβίωση ειρήνη και σταθερότητα για το Ισραήλ σε κανένα διεθνή φορέα και οργανισμό. ήταν τα πράγματα δεδομένα, βεβαίω θα μπορούσαμε ο καθένα να εκφράσουμε τι κατηγορίε και τι καταγγελίε μα. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κράτο το οποίο έχει την πολυτέλεια να καταπιέζει του ε, πολίτε του. Και μπορεί ο κύριο Σάιτ να ήταν κάπω πιο μετριοπαθή από ότι άλλοι ομιλητέ αργότερα. Αλλά πάντω αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν να διαπραγματεύονται σοβαρά απέναντι στο Ισραήλ δεν έχουν δεδομένα αυτά δεν έχουν ως δεδομένες αυτές τις πεπιθήσεις, ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακούσατε από την ε, παρουσίαση της έκθεσης Gladstone, ούτε και ισχύει το γεγονός, αφού όλοι ακούσαμε τα όσα λέει ο ε, πρεσβευτής ε, του Ισραήλ, ότι δηλαδή δεν χρησιμοποιεί το Ισραήλ τον όρο τρομοκράτα για κάθε είδου άμαχο πολίτη. Δεν μπορούμε εμεί λοιπόν να θέτουμε το Ισραήλ στο εδόλο του κατηγορούμενου και αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τα πράγματα άσπρα μαύρα, ούτε είναι οι φίλοι μα οι Ισραηλοί λόγω τη θρησκευτική του προσέγγιση, ούτε φίλοι μα οι μουσουλμάνοι επειδή είναι μουσουλμάνοι. Είναι ε, δεδομένες μόνο οι ευθύνες μας ως βουλευτών λόγω του ε, λειτουργήματος το οποίο επιτελούμε και πρέπει να συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό τον επικοδομητικό στο διάλογο γιατί είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να δούμε το σφαιρικά τον διάλογο αυτό και είναι ευθύνη σας κυρία Πρόεδρε πιστεύω γιατί βεβαίως ήταν πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον το ότι οργανώσατε τη συζήτηση σήμερα αλλά και για το μέλλον θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, σοβαροί προς το να προσδιορίσουμε το, τα θέματα στα οποία μπορούμε να συμβάλλουμε επικοδομητικά. Εγώ βεβαίω ε, θεωρώ ότι ο κάθε ένας από τους βουλευτές εδώ έρχεται καλόπιστα να προσφέρει και να συμβάλλει στην ειρήνη. Το να λέμε όμως οι Ισραηλινοί δεν θέλουν την ε, ειρήνη, δεν θέλουν τη διαπραγμάτευση κτλ. Δεν μπορεί να ισχύει και εγώ θα φυλαχθώ και δεν πρόκειται να το πω αυτό ποτέ για κανέναν από τους άλλους εδώ παριστάμενους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να κοιτάξουμε από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε εδώ πέρα και, για τα, θέματα, και τα θέματα της ενότητας των Παλαιστινίων και την προόδο αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε πολύ καλά όταν καθοριστικά τα γεγονότα της Γάζας, ξέρετε πολύ καλά ότι για τη συνέχεια χρειάζεται ο συνομιλητή και προσπαθείτε να εξασφαλίσετε αυτόν τον συνομιλητή από πλευρά Παλαιστινίων. Πού βρίσκεται λοιπόν η ενότητα η εθνική των ε, ε, Παλαιστινίων. Και θα ήθελα να ακούσουμε και από τον κύριο Σαΐτ κάποιες απαντήσεις στην υπόθεση αυτή. Ερωτώ λοιπόν εδώ εάν μπορούμε να συμβάλλουμε επικοδομητικά στη συζήτηση. Γιατί άμα είναι να καταγγέλουμε ο ένας τον άλλον μόνο και να ε, κάνουμε δίκες προθέσεων, ε, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θέματα του, των υδάτινων πόρων βεβαίω και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εάν λοιπόν μπορούμε με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε επικοδομητικά, με τρόπο μετριοπαθή, σεμνό και ταπεινό, τότε ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Διαφορετικά μπορούμε να κινδυνεύσουμε να δούμε μια κρίση σαν αυτή να συνεχίζεται επαόριστον. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο στον επόμενο μιλτή. Κύριε Αλφετή, θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στους ομιλητέ που ανέφερα πριν και εσεί θα έχετε το λόγο εν συνεχεία. Ο κύριος Βέρλα από τη Μάλτα. Ευχαριστώ. Όπως σε αντίστοιχε συναντήσει, μετά από τον τέταρτο ή πέμπτο ομιλητή, ε, έχουν καλυφθεί όλα τα θέματα. Ε, ε, επειδή εγώ δεν θα μπορέσω να τα πω καλύτερα από όσα τα είπε η κυρία Φλότ. Ε, δεν θα μακρηγορήσω. Ο, αμέσως πριν από την συζήτηση, ο πρέσβης είπε ότι υπάρχει μια επιθυμία να επιτεθείτε στο Ισραήλ και να το βάλετε στη γωνία. Θεωρώ ότι είμαι ένας από αυτούς που δεν είμαι υπέρ του Ισραήλ, ούτε ε, και υπέρ του, των Παλαιστινίων. Είμαι υπέρ της ειρήνης. Δυστυχώ όμως πρέπει να θέσουμε ερωτήσει προς τους Ισραηλινούς. Δεν ξέρω αν θέλω να το χαρακτηρίσω ε, ευκαιρία ή ατυχία, αλλά είχα την ε, ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, ε, μία φορά αμέσω μετά την στρατιωτική επίθεση να επισκεφθώ τη Γάζα και αμέσω μετά και μια δεύτερη φορά το Μάιο. Οι μνήμε αυτές που μου δημιουργήθηκαν δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι σήμερα, σε αυτόν τον αιώνα, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είναι κυριολεκτικά ε, δέσμοι σε μια ανοιχτή φυλακή. Πήγαμε στα στρατόπεδα, πήγαμε στο, μιλήσαμε με τον λαό, ζουν σε άθλιες, σε μίζερες συνθήκες και αυτή η κατάσταση με τίποτα δεν δικαιολογείται. Θα ήθελα τώρα να εστιάσω σε ένα μόνο πράγμα. Ακούστηκαν πολλά. Εγώ θέλω να μιλήσω για, ε, για τους επικισμούς και μόνο. Μπορεί να είμαι απλουστευτικός και σχηματικός. Το 1982 μεταξύ του Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι ε, και του Μωσέ Νταϊάν, τότε ο Μπούτρος Γκάλι ήταν ε, υπουργός εξωτερικών της ε, Αιγύπτου, είχε τεθεί αυτό το θέμα των επικισμών. Είχαν πει τότε ότι είναι το κρίσιμο θέμα. Και εξακολουθεί να είναι και σήμερα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Δηλαδή, αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Γιατί είναι τόσο απαραίτητοι οι επικισμοί. Είναι μια δήλωση. Στην Ανάπολη το Ισραήλ δεσμεύτηκε να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών. Δεν το έκανε όμως. Δεν υπάρχει χώρο στο Ισραήλ για να ε, ζήσουν και να εγκατασταθούν νέε Ισραηλινές οικογένειε. Ή είναι οι ίδιες οι Ισραηλινές οικογένειες που θέλουν να εγκατασταθούν όχι στο Ισραήλ, στην επικράτεια του Ισραήλ, αλλά στα κατεχόμενα. Είναι τόσο μεγάλος ο πληθυσμός που σας χρειάζονται οι επικισμοί δεν αναγνωρίζει το γεγονό ότι με βάση το διεθνέ δίκαιο δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου επικισμοί σε κατεχόμενα εδάφη υπό την Σύμβαση της Γενέβης. Αυτό είναι το, εν, το, το πιο κρίσιμο θέμα, το θέμα των επικισμών. Τελικά τι να πω, ότι δεν χρειάζονται την ειρήνη οι Ισραηλινοί, αφού ζουν με αυτές τις συνθήκες. Γιατί χρειάζεστε αυτή τη διαδικασία. Θέλετε να εκφράσετε την ανωτερότητά σας απέναντι στους Παλαιστινίους ή να εκφράσετε την πλήρη αδιαφορία για τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και την διεθνή κοινή γνώμη. Είναι πολιτική δήλωση. Και πραγματικά ε, αισθάνομαι άσχημα που το θέτω έτσι. Είναι ένας εύσχημος τρόπος για να καθυστερήσετε την προσέγγιση Ισραηλινών και Παλαιστινίων τη στιγμή που κατέχετε και προσαρτάτε τα παλαιστινιακά εδάφη, δεν αφήνεται γη στους Παλαιστίνιους, δεν αφήνεται τίποτα για να διαπραγματευθείτε. Στην πραγματικότητα, εκ των πραγμάτων, απομακρύνεται από αυτή τη διαδικασία τους Παλαιστίνιους. Είναι αποτελεσματική αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Βέλλα. Ο κύριος Χατζηνικολά από την Κύπρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πολύ σύντομος γιατί είναι θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει επανελειμμένα σε αυτή την Επιτροπή και πάντοτε σε αυτές τις συζητήσεις καταλήγουμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που πιστεύω αυτό το κοινό σημείο δεν είναι μόνο εμείς εδώ που καταλήγουμε αλλά αν κάναμε ένα δημοψήφισμα μεταξύ των λαών ολόκληρης της περιοχής, ιδιαίτερα της νοτιοανατολικής Μεσογείου το 100% θα ψήφιζαν ότι να είμαστε όλοι υπέρ τη ειρήνη. Για να επικρατήσει όμω αυτή η ειρήνη, ε, χρειάζονται αρκετέ προσπάθειε από όλου μα. Και νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή, η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερικανική Κυβέρνηση, όλοι, εν πάση περιπτώσει, όσοι εμπλέκονται σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει όλοι να αναπτύξουν πρωτοβουλίε. Είναι απαράδεκτο, και το τονίζω αυτό, να επικρατεί σήμερα το δίκαιο του ισχυρού σε αυτόν τον αιώνα που ε, με όλες αυτές τις κατακτήσεις που έχουν οι λαοί και δυστυχώς να επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού αντί να επικρατεί το διεθνές δίκαιο. Στην περιοχή σίγουρα υπάρχει το πρόβλημα με τους ε, επικισμούς, με τον πόλεμο στην Γάζα, όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως είναι και έχουμε πει όλες τις εμπειρίες τις οποίες έχουμε ζήσει. Ναι, έχουμε πάει στη Γάζα, έχουμε πάει και στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006, και δεν θα ήθελα ούτε ε, να πω ούτε τέλο πάντων τι εμπειρίε που ζήσαμε ο καθένα, γιατί ο πόλεμο είναι παντού πόλεμο. Είτε είναι στη Γάζα, είτε είναι στο Ιράκ, είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι ξέρω εγώ οπουδήποτε. Ο πόλεμο αυτά φέρνει. Και δεν είναι πολέμοι μεταξύ των λαών. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν λαοί που θέλουν να κάνουν πολέμου. Είναι τα στρατηγικά συμφέροντα του κάθε ε, κάθε κράτου, εν πάση περιπτώσει, τη κάθε κυβέρνηση, στι συγκεκριμένε συνθήκε. Ε, εγώ επιμένω στην πρόταση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες. Και οι πρωτοβουλίες αυτές δεν είναι απαραίτητα να κατευθύνονται προς τις κυβερνήσεις. Ναι, να απευθύνονται στις κυβερνήσεις, αλλά υπάρχουν και μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις. Υπάρχουν τέλο πάντων χίλια δυο άλλα ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε κι εμείς έτσι που να δημιουργήσουμε τουλάχιστον έναν κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών των λαών, μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Όπω για παράδειγμα μπορεί να είναι το περιβάλλον, μπορεί να είναι το νερό, μπορεί να είναι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, μπορεί να είναι οικονομία, μπορεί να είναι πολιτισμό. Υπάρχουν χίλιοι δυο τομεί που μπορούμε να αναπτύξουμε συνεργασίε στο να καταφέρουμε και να επιβάλλουμε αυτό το οποίο πρέπει να επιβληθεί ιδιαίτερα σε αυτήν την δύσκολη, αυτήν την ταλαιπωρημένη περιοχή. Έχω ακούσει με προσοχή την αντιπρόσωπο τη Τουρκία, η οποία μου είναι και πολύ συμπαθή. Ε, έχουμε ξανασυναντηθεί και σε άλλα συνεδρία. Ναι, η Τουρκία σήμερα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. Ε, Έχουμε ζήσει τον πόλεμο και στην ίδια την Κύπρο δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτέ τι εμπειρίε. Όμω η Τουρκία έχει υποχρέωση σήμερα, αντί να δίνει ευχέ να επιληθεί το Μεσανατολικών, έχει υποχρέωση να βοηθήσει στον και των Κυπριακών. Υπάρχουν συνομιλίε στην Κύπρο σήμερα και το κλειδί αυτή τη λύση σίγουρα είναι στην Άγκυρα. Εμεί, σαν Κύπρο, στηρίζουμε την προσπάθεια τη Τουρκία και ναι, να γίνει ευρωπαϊκό κράτο η Τουρκία. Και έχει όλα τα χέγγια. Με την προπόθεση όμω ότι και αυτή θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Εγώ τελειώνοντας, ε, έχω αρκετά σίγουρα άλλα να πω αγαπητοί πρόεδρος, αλλά θα συμβαστώ το χρόνο, θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο. Τελευταία έχει απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ στον ε, πρόεδρο της, Αμερική, Αμερικής, τον κύριο Ομπάμα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, ας ελπίσουμε ότι αυτό το βραβείο Νόμπελ θα λειτουργήσει ως πηξίδα για τον ίδιο και την Αμερικάνικη κυβέρνηση, έτσι που να εξεύρουμε την πραγματική ειρήνη και τη συνεργασία και την πρόοδο σε όλα τα μήκη και πλάι του πλανήτη. Αυτόν το βραβείο Νόμπελ ας βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε και να κρατήσουμε το διεθνές δίκαιο, να επιβληθεί η ειρήνη και όχι το δίκαιο του ισχυρού που υπάρχει σήμερα. Ε, θα μείνω μέχρι εδώ γιατί υπάρχουν σίγουρα και άλλα ζητήματα που θέλω να σχολιάσω, όμως σε επόμενο χρόνο θα μείνω μέχρι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάει ο καιρό, ο κύριο Πρέσβη πρέπει να εγκαταλείψει το βήμα σε λίγο, οπότε θα δώσω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Ελφακή. Ένα λεπτό, ε? Ένα λεπτό. Να θέλω κι εγώ να έχω. Ο πρέσβης πρέπει να φύγει, γι' αυτό. Ναι, ναι, θέλω λιγάκι να του ξαναθυμίσω μερικά πράγματα πριν αποχωρήσει την ε, μέρα της ε, κατανομής στο Συμβούλιο Ασφαλείας είχε αναφερθεί ότι είναι εβραϊκό κράτος. Ο τέος ο Υπουργός Τρούμαν τότε ήταν εκείνος ο οποίος το διέγραψε αυτό και είπε ότι είναι το κράτο του Ισραήλ, από την έκανε άλλη μεριά ένα Παλαιστινιακό κράτο. Αυτό το πρώτο. Δεύτερον, κάθε φορά που μιλάνε για εβραϊκό κράτο, αυτό δίνει έναν λόγο ύπαρξη παραπάνω στου ακραίου μουσουλμάνους να μιλάνε για μουσουλμανικό κράτος. Οπότε τελικά καταλήγουμε σε μια θρησκευτική αντιπαράθεση και όχι πολιτική αντιπαράθεση, κάτι που επίσης υπονομεύει τις δυνατότητες και τις ειρηνευτικές προσπάθειες που γίνονται και, μας, ε, και οδηγούν τους Παλαιστινίους σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Έπειτα οι Παλαιστίνοι στο Ισραήλ είναι σαν δεύτερης κατηγορίας ε, πολίτες, αυτόματα. Αν λοιπόν θέλετε να αναγνωρίσετε τη λύση των δύο κρατών και να μιλάτε γι' αυτό αλλά χωρίς πραγματικές προσπάθειες, τότε να μιλάμε για δημοκρατικό κράτος, για λαϊκό κράτος, κοσμικό κράτος, που να είναι μέσα και οι Παλαιστίνοι, οι Άραβες, οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι, αλλά αυτό το απορρίπτετε εσείς. Οπότε μην μιλάτε για εβραϊκό κράτος, γιατί αυτό δεν σας συμφέρει τελικά. Επίσης θέλω να επιθυμίσω στον πρέσβη ότι το όνομά σα είναι γνωστής οικογένεια Ισραηλινών, γνωστών πολιτικών και νομίζω ότι αυτό πρέπει να σα θυμίσει πόσο μεγάλη ε, ανοχή δείχναμε εμείς πριν από μερικά χρόνια. Ο πρέσβης να απαντήσει. I <clears throat> want to thank Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, εκπρόσωπο από την Αίγυπτο για τα καλά του λόγια. Έχετε δίκιο για αυτά που είπατε για το Κάιρο. Ήμουνα μια φορά στη συναγωγή. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες οικογένειες. Ε, θα θυμάστε ότι ο Ανρί Κουριέλ, που είναι από την οικογένειά μου, δολοφονέθηκε στην, στο Παρίσι. Αλλά δεν θα πρέπει να μπούμε τώρα σε παράθεση γεγονότων. Αν πάτε στο ψήφισμα του ΟΗΕ, θα δείτε ότι το 47 υπόθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα Ισραηλινό κράτος και ένα Αραβικό κράτος, όχι μουσουλμανικό κράτος. Έτσι, η λύση είναι δύο κράτη, κρατική λύση λοιπόν. Εμείς δεν, θέλουμε χρειαζόμαστε την αναγνώριση κανενός. Ε, δεν θέλουμε να μας αναγνωρίσει τον εθνικό μας χαρακτήρα. Το ΕΙΠΑ, γιατί. Γιατί ακόμα υπάρχει στην Ισραηλινή κοινή γνώμη αυτό το αγκάθι για το αν υπάρχει αναγνώριση του Ισραήλ. Όσο έχει. Αυτό τι σημαίνει. Με τον εθνικό του χαρακτήρα. Με όλα τα χαρακτηριστικά του. Και δεν είναι ίσονο σημασία θέμα αυτό, γιατί αφορά τον πυρήνα της λύσης, την ουσία της λύσης, την ουσία του προβλήματος. Κάτι άλλο το οποίο είναι αντίρρητο είναι ότι με το να λέμε νούμερα η Συριακή ας πούμε αντιπροσωπεία είπε ότι οι επικισμοί είναι το 15% της επικράτειάς μας. Ε, νούμερα έτσι, αριθμητικά στοιχεία. Αν δεν κάνω λάθος, θα το κοιτάξω βέβαια. Νομίζω ότι δεν είναι 15%, είναι 1,5%. Ε, είναι πολύ παρακάτω από το 15% λοιπόν. Πριν ε, έρχεστε εδώ στο και μιλάτε για τέτοια νούμερα, τέτοια ποσοστά, σας παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία σας. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και είναι θετικό και που δεν το συζητήσαμε αυτές τις μέρες είναι η βελτίωση στη δυτική όχθη τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, από την εποχή που ήρθε στην ε, εξουσία η κυβέρνηση Νετανιάχου, νομίζω ότι υπήρχε μια πολύ έντονη βελτίωση στην κατάσταση στη Δυτική Όχθη και δεν νομίζω ότι η εκπρόσωπο τη Παλαιστίνη θα το αμφισβητήσει. Δεν λέμε ότι αυτό έγινε χάρη στο Ισραήλ, ίσω ε, και χάρη στη διαχείριση των ε, Παλαιστινίων και στη διεθνή βοήθεια, αλλά και χάρη στα βήματα που έχει προωθήσει το Ισραήλ, έρει τα οδοφράγματα. Κάνει κινήσεις, τις οποίες δεν θα πρέπει να τις ε, ξεχνάμε. Νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχουν καλά νέα από τη Δυτική Όχθη. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Γιατί μιλάμε για μια διαδικασία οικοδόμησης κράτους, που είναι πολύ σημαντική, αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη δικρατική λύση. Ε, έχετε την έκθεση Goldstone. Την έχετε στους φάκελούς σας, από ό,τι άκουσα που μιλάει για την Ισραηλινή απόκριση. Έχουμε πρόβλημα με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και δεν είμαστε οι μόνοι που έχουν πρόβλημα με το Συμβούλιο. Είναι ένα Συμβούλιο που η πλειοψηφία των κρατών δεν προωθούν, εκεί μέσα δεν προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια πολιτική έκθεση αυτή που έχει κάνει το Συμβούλιο. Θέλω να υπενθυμίσω στην Προεδρία ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστήριξαν την εντολή της ε, Επιτροπής Goldstone και δεν υποστήριξαν ε, το ψήφισμα που πρόσφατα υιοθετήθηκε στη Γενέβη. Α μην σα μιλήσω για κάθε παράγραφο τη ε, έκθεση και για κάθε πρόβλημα που έχει η έκθεση, αλλά υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα που δεν αφορούν μόνο το Ισραήλ στην έκθεση αυτή, αλλά την αρχή του δημοκρατικού κράτους που δρά για λόγους αυτοάμυνας. Ε, το Ισραήλ παίρνει ρίσκα για την ειρήνη. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την ασφάλειά του. Όταν κάνουμε αυτές τις συζητήσεις λοιπόν δεν θα πρέπει να λησμονούμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ όλους. Ζητώ συγγνώμη που πρέπει να φύγω. Υπάρχουν και άλλα θέματα στη Μέση Ανατολή, βεβαίω, τα οποία πρέπει να συζητηθούν και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη Μεσόγειο. Σα ευχαριστώ για την υπομονή σα και σα ευχαριστώ όλου ιδιαίτερω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη, για την παρουσία σα σήμερα το πρωί. Γνωρίζεστε. Μάλιστα. Θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους κύριους ομιλητές. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, γεια σας. Η κυρία Σαγίτ έχει φύγει, ο κύριος Αμπταλά θα πάρει τώρα το λόγο και θα μιλήσει ανταυτής. Εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στην κυρία Κέρντιν και εν συνεχεία τελευταίο στον κύριο Ρίπεκ για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Κύριος Αμπταλά. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέρφους από διάφορα κοινοβούλια. Κοιτάξτε, στη δικιά μας την παράδοση, παρόλο που έφυγε ο πρέσβης, αλλά αν κάποιος σας χαιρετήσει με έναν τρόπο, πρέπει να ανταποκριθείτε εσείς με έναν ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει ένα βήμα προς το μέρος σας, εσείς κάνετε δύο βήματα προς το μέρος του. Αυτή είναι η παράδοση, συνήθεια. Πολλά θέματα έχουν συζητηθεί εδώ. Και πριν είχαν λάβει χώρα για τα ίδια θέματα και άλλες συζητήσεις, πολλές πολλές. Ένα έχει αλλάξει. Νέες παραβιάσεις του νόμου από την ίδια πλευρά. Που βρίσκεται, αν όχι σε πλήρη απομόνωση, στην μειοψηφία. Δεν μας εκπλήσει. Εδώ όμως πρέπει να φροντίζουμε για την προστασία του διεθνούς δικαίου, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα, πυλώνες. Οι κοινοβουλευτικοί τα θεωρούν πολύ σημαντικά και τα σέβονται. Τώρα όμως νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα ακόμα προς τα προς Δράση. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να αποφύγουμε την επόμενη φορά να συζητάμε περίπου τα ίδια πράγματα συν άλλη μια παραβίαση, επίθεση, κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, στα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ και συζητήθηκαν, θέλω να προσπαθήσω να διευκρινίσω κάποια. Το πρώτο και το πιο εύκολο είναι ο εβραϊκός χαρακτήρας του κράτους του Ισραήλ. Αυτός ο εβραϊκός χαρακτήρας είναι κάτι που ποτέ δεν ζήτησε η Αίγυπτος όταν υπογράφηκε η αμοιβαία αναγνώριση το 1979. Κανείς δεν το ζήτησε από την Ιορδανία όταν υπέγραφε η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία το 1994. Κανείς από τα Ηνωμένα Έθνη. Τίθεται μόνο επειδή υπάρχει θέμα μεταφοράς των Αράβων Παλαιστινίων που είναι Ισραηλινοί υπήκοοι που έμειναν εκεί και θέλουν να τους διώξουν εκτός συνόρων. Γι' αυτό τίθεται αυτό το ζήτημα. Υπάρχει λοιπόν ε, μεγάλη υποψή, όπως καταλαβαίνετε γιατί θέλει να βάλει αυτή τη νέα προϋπόθεση όσον αφορά την αμοιβή αναγνώριση ενώ το PLO, η Οργάνωση για την Απευθύνση της Παλαιστίνης όταν συζητούσε αυτά, ήξερε ότι ποτέ δεν είχε ζητηθεί από το Ισραήλ να αναγνωριστεί σαν εβραϊκό κράτο. Τώρα ζητάνε κάτι παραπάνω λοιπόν. Κάποιος από τους ομιλητέ είπε ότι ο μόνος στόχος, γιατί το κάνουν αυτό δηλαδή, είναι για να καθυστερήσει ή οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους. Είναι μια πολιτική απόφαση που παίρνει το Ισραήλ, το οποίο πρέπει να δεχτεί τα δύο κράτη. Και όταν ο κύριος Νιατανάου τόνισε την λύση δύο κράτη, γιατί αυτό το βασικό στοιχείο της νέας Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε Παλαιστινιακό κράτος που να μην ελέγχει ούτε τον αέριο χώρο, ούτε τα σύνορα, ούτε την Ιερουσαλήμ, να μην έχει δικαίωμα στρατιωτικής δύναμης και τέτοια. Βασικά περιέγραφε ένα κράτος το οποίο να είναι υπό την κυδαιμονία των Ισραηλινών. Λοιπόν, διαπραγματεύσεις. Εμείς ποτέ δεν απορρίψαμε τις διαπραγματεύσεις. Συμφωνούμε. Αν υπάρχει μια σύγκρουση, προφανώς και χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε κάπου. Όμως οι διαπραγματεύσεις αυτές από τη δικιά μας την εμπειρία ξεκίνησαν στη Μαδρίτη. Μετά είχαμε Ουάσιγκτον. Μετά είχαμε διάφορες επιτροπές, διμερείς. Οι διαπραγματεύσεις όμως δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι το μέσο για να πετύχουμε την ειρήνευση. Όμως στις διαπραγματεύσεις αυτές διαπιστώσαμε ότι το Ισραήλ εντωμεταξύ αύξανε τις... ε, τους επικισμούς. Από το 1991 μέχρι τώρα έχει αυξήσει τους επικισμούς από 70 σε σχεδόν 400 σήμερα. 112 από αυτούς ήταν ε, ουσιαστικά παράνομοι επικισμοί όχι μόνο απέναντι στο διεθνέ δίκαιο, αλλά και απέναντι στο ίδιο το Ισραηλινό δίκαιο. Όμως ποτέ δεν ελήφθησαν κυρώσει, ποτέ δεν ζήτησε η Αμερική, η Ευρώπη αυτοί οι επικισμοί να καταστραφούν, οι οποίοι έγιναν μετά το Μάρτιο του 2001. Οι δε επικοί αυξάνονται βέβαια. Από 100.000 σε περίπου 500.000 σήμερα. Το τείχος επίσης που χωρίζει με apartheid που χωρίζει τους Παλαιστινίους από τους Παλαιστινίους δημιουργήθηκε μέσα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τι τις έχουμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις αν χρησιμοποιούνται μόνο για να ε, είναι σαν άλοθη για το Ισραήλ για να κάνει ό,τι θέλει. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Παλαιστινίους και το Ισραήλ πρέπει να είναι υγιή, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, που λέμε να πάμε στα σύνορα του 67. Ο Μπούς βέβαια έλεγε της ε, Κεχηρίας που να είναι αυτή που χωρίζει τους Ελληνούς από τους Παλαινιστίους. Ωραία. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν πρέπει να χρησιμεύουν για να προστατευτεί η γη. Να μην επιτραπεί δηλαδή καμία περίπτωση νέου επικισμού. Ενώ, παρόλο που το έχει πει και ο κύριος Μίτσελ και έχει ξεκινήσει η έκθεση το, από το 2001, προσπαθούν να λύσουν αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά τους επικισμούς λοιπόν, είναι αλήθεια ότι το μέγεθος που επιτρέπει 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι, λέει η Συμφωνία του Όσλο γι' αυτό. Όμως οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν επεκτείνει και ακόμα και σε περίπτωση πάνω από 50. Και έτσι κανένας Παλαιστίνιος δεν μπορεί να πλησιάσει τους επικισμούς αυτούς, που είναι το 15% είπαμε τώρα της γης. Και έτσι προστίθεται στα κατεχόμενα και αυτή η γη. Οι επικισμοί όμως είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν είχε τεθεί στους προηγούμενους, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Ούτε οι Αμερικανοί έλεγαν την αλήθεια. Εμείς περιμένουμε οι Αμερικανοί να ψωθούν και να πούνε έγινε λάθος. Έπειτα, ο δικός χάρτης. Η πρώτη εκδοχή έβαλε υποχρώσεις και στις δύο πλευρές. Η πρώτη από τις υποχρώσεις για το Ισραήλ ήταν να σταματήσει την επέκταση των επικισμών. Στην Ανάπολη. Νοέμβριος 2007. Επίσης συμφωνήθηκε και οι Αμερικανοί ήταν εκείνοι που το πρότειναν να σταματήσουν όλες οι δραστηριότητες επικισμού ποτέ στο παρελθόν δεν μπαίνανε. Ε, να, μπήκανε. Αλλά οι Ισραηλινοί δεν το δέχονται σαν σημείο αναφορά για παρετέρω διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί να συζητάμε 60-80 χρόνια για τίποτα. Και από το Σαμίρ έχουμε μάθει διαπραγματεύσεις χωρίς να δίνουμε τίποτα. Δεν γίνεται. Ναι, θα είμαι σύντομος. Πάντως, ας προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε δράση και όχι να μιλάμε και να μιλάμε και να μιλάμε. Φυσικά και έχουμε λόγο. Ερωτήματα. Γιατί Ευρώπη. Μερικές ευρωπαϊκές χώρες χτίζουν την εξωτερική τους πολιτική πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά την έκθεση Goldwood ορισμένοι κατέληψαν την αίθουσα για να μην συμμετάσχουν ακριβώς στην ψηφοφορία και άλλοι κράτησαν θέση αποχής. Μα δεν είναι συμβατό αυτό με τις αρχές τις οποίες λένε ότι βασίζουν την πολιτική τους. Ελπίζουμε οι Αμερικανοί να μην επιτρέψουν στους αυτούς τους να παραπλανηθούν από τους Ισραήλ για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Merci. Donc je donne la... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Κέρσλιν. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη. Καταρχά ευχαριστώ τους ομιλητές εκείνου οι οποίοι αναφέρθηκαν στο βραβείο Νόμπελ που απενεμήθη στον πρόεδρο Ομπάμα. Ασφαλώς θα αντιλαμβάνεστε ότι το εκλαμβάνει περισσότερο σαν πρόκληση τη δουλειά δηλαδή που έχει να επιτελέσει περισσότερο παρά επιβράβευση κάποιας δουλειάς που έχει γίνει. Είπε ο ίδιος ότι αισθάνεται ε, μεγάλο το βάρος της ευθύνης από την ε, απονομή αυτού του βραβείου. Ο μιλητή από την Ισία αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα. Η Τινησία ασφαλώ έχει διαδραματίσει ρόλο επικοδομητικό, έχει συμβάλει πολύ στην ειρηνευτική διαδικασία και υπολογίζουμε θα στοιχιστεί αυτή η βοήθεια όχι μόνο από τα κύρια κράτη, ε, τα κύρια παρόντα στην περιοχή επικράτη, αλλά και από όλα τα κράτη και της Ευρώπης και της περιοχής ευρύτερα. Επίσης, υπόθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει συνάντηση στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο, ε, πράγμα το οποίο οδήγησε τελικά σε παρουσίαση ενός σχεδίου. Υπήρχε η ελπίδα, πιστεύουμε, ότι θα διεξαγόταν αυτή η συνάντηση μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά δεν θα χαρακτήριζα την μη διεξαγωγή της συνάντησης αυτής ως αποτυχία. Ο κύριος Μίτσελ ο ίδιος είπε μάλιστα όταν ανέλαβε καθήκοντα όταν ανακοινώθηκε ο διορισμό του καλύτερα, ότι σε σχέση τέλο πάντων με την Ιρλανδία και τι προσπάθειέ του εκεί, χωρί να θυμάμαι επαρκώς, ε, επακριβώ τον αριθμό των ημερών που ανέφερε, είχε πει ότι ε, είχε περάσει από 800 τόσε μέρε αποτυχία πριν φτάσει στη μία μέρα επιτυχία στι διαπραγματεύσει. Αυτό είπε ο κύριο Μίτσελ και πιστεύω ότι συνεχίζει την προσπάθεια αυτή και ε, στην υπόθεση του Ισραήλ. Ο κύριο Σταμπάκη νομίζω είπε επίση ότι θα πρέπει τα Ηνωμένε Πολιτείε να εμπλακούν περισσότερο στην ε, συμφιλίωση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ούτε θα πρέπει όμω ούτε θα ήθελαν ασφαλώ να είναι η μόνη χώρα η οποία προβάλλει τα θέματα αυτά. Εμεί υποστηρίζουμε και τι προσπάθειε τη Αιγύπτου για την συμφιλίωση μεταξύ Παλαιστινίων. Ε, πολύ δύσκολο έργο ασφαλώ. Και θα συνεχίσουμε να του υποστηρίζουμε. Είναι μια προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να συμβάλλουν πολύ. Θα σα παραπέμπω επίσης ότι θεωρώ ότι θα ήταν ε, χρήσιμο ε, στις δηλώσεις της ε, Υπουργού των Εξωτερικών κυρίας Κλίντον όπου καταγράφει μετά τη συνάντησή τη με τον Πρωθυπουργό Νατανιάχου και δηλώνει η κυρία Κλίντον, επαναλαμβάνοντα τα έχει πει και ο, ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι δεν είναι αποδεκτή η συνέχιση των επικισμών των Ισραηλινών. Δηλώνεται η κυρία Κλίντον και παραθέτω ότι το Ισραήλ δεν έχει συγκρατήσει τους επικισμούς, δηλαδή δεν ικανοποιεί τις ε, αμερικανικές προτιμήσεις. Όμως θα ήθελε, συνεχίζει, να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για ειρήνευση ή προόδο τέλο πάντων στη σχέση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Πιστεύουμε ότι ίσως θα ήταν ε, Ίσως πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να ξεκινήσουν και πάλι οι έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο στόχος των δύο κρατών και νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, να ομολογήσουμε ότι οι συνεχιζόμενοι επικισμοί αποτελούν πρόσκομα στην πρόοδο. Θα σταματήσω όμως γιατί ξέρω ότι όλοι μπορούμε να μιλήσουμε για πολλή ώρα αλλά εν πάση ευχαριστώ πολύ να αφήσω το λόγο και στους άλλους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κέρτιν. Κύρια Ρίτζιμπερκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να εξηγήσω τη θέση και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάλυση που κάνουμε για την κατάσταση της ε, διαδικασίας της Μέσης Ανατολής και να απαντήσω σε ερωτήσεις ε, που θέσατε. Δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα όσα έχω ήδη πει. Θα ήθελα απλώς να συνοψίσω τη θέση μας ε, σε τρία πολύ σύντομα σημεία. Θα θέλαμε να γίνουν διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα, τα, τα τελικά, τα σημαντικά. Θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση εκ του σύνεγγης, ιδίως στη Γάζα και την Ιερουσαλήμ. Θα το κάνουμε βασιζόμενοι στην ε, στεναρή μας δέσμευση ότι το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να είναι η προϋπόθεση και η βάση για μια λύση στην ε, Άραβο-Ισραηλινή σύγκρουση. Και τρίτον, θα συνεισφέρουμε όσο πιο ενεργά μπορούμε, καθώς θα ε, συνεργαζόμαστε και θα προωθούμε την ε, εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με όλους τους υπόλοιπους φίλους μας στην περιοχή. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω τον απόντα φίλο μου, τον ε, πρέσβη Κουριέλ και την εκπρόσωπο Σαχίντ, την Αμερικανίδα εκπρόσωπο, εσάς κυρία Πρόεδρε και βεβαίως τους ε, εκπροσώπους από τα διάφορα κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ρίτμπεργκ. Τώρα θα δώσω στον κύριο Ντελπικά, τον αντιπρόεδρο της ε, συνέλευσης, το λόγο για να κλείσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε, είμαι στην Επιτροπή αυτή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και παρακολουθώ τις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής, ακόμα πιο πολύ το ξέρει και το Μισελ Μπλό, είναι πάρα πολύ καιρό που ασχολούμαι με αυτά. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία συζήτηση ίσως την πιο ενδιαφέρουσα. Και γιατί? Γιατί εκατέρωθεν, έτσι έχουμε ζήσει πολύ έντονη συζητήσει και στην Αθήνα και αλλού, αλλά αυτή τη φορά βγαίνει κάτι θετικό και από τις δύο πλευρές οφείλεται στους συμμετέχοντες και τους ευχαριστώ και στον πρέσβη και στην κυρία. Νομίζω λοιπόν ότι προχωράμε προς μια καλή κατεύθυνση. Δύο λόγια όμως, πολύ απλά. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, ενώ η Επιτροπή μας. Γιατί, ναι, διαχωρισμός εξουσίας, νομοθετική από τη μια, εκτελεστική από την άλλη. Εμείς δεν είμαστε εκτελεστικοί, εμείς είμαστε η νομοθετική εξουσία. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να προχωρήσουν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το είπαν όλοι εδώ, όλοι είναι για την ειρήνη, οπότε κανένας δεν τα βάζει με κανέναν εδώ ε, σήμερα. Εγώ είμαι παιδί της γερμανογαλλικής συμφιλίωσης. Ξέρω τι πάει να πει συμφιλίωση. Βέβαια αυτά έγιναν παλιότερα. Διάλογος, ε, διαπραγματεύσεις, έφραυστη ειρήνη στην αρχή, αλλά σιγά σιγά θα υπάρξει, τουλάχιστον ελπίζουμε ότι θα υπάρξει αυτή η ειρήνη. Εμείς οι κοινοβουλευτικοί όμως που είμαστε πολιτικοί, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Δεν έχουμε την εξουσία να πάρουμε αποφάσεις, έχουμε όμως τη δύναμη να επηρεάσουμε τα πράγματα ως κοινοβούλιο, να επηρεάσουμε ίσως τις κυβερνήσεις μας, τους διπλωμάτες μας. Έχουμε όμω και τη δύναμη να επηρεάσουμε την κοινή γνώμη προ τη σωστή κατεύθυνση. Και αναρωτιέμαι, κυρία Πρόεδρε, μήπω το σώμα αυτό δεν θα έπρεπε κάποια μέρα να αποφασίσει αλλά όχι όπω συνήθω κάνουμε ψηφίσματα με 42 σημεία, 1, 2, 3, 4, θέλουμε αυτό, και εκείνο το άλλο. Όχι, αυτά να τα ξεχάσουμε. Δεν βοηθάνε εξάλλου και κανένα δεν το αρνείται αυτό. Δεν έχουν βοηθήσει. Λοιπόν, όλα μπορεί να είναι σωστά, καλά. Σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, αλλά κανένα δεν τα διαβάζει από την αρχή μέχρι το τέλο. Οπότε, μήπω η Επιτροπή μα, κυρία Πρόεδρε, θα έπρεπε καλύτερα να δουλέψει πάνω σε ένα μικρό κείμενο, το οποίο να είναι κείμενο που να προκαλεί λιγάκι αντιδράσεις από την κοινή γνώμη. Λέγοντας, ναι, υπάρχουν βουλευτές από το Βορρά και από το Νότο που συμφωνούν μεταξύ τους για να έχουμε ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω τι γνώμη έχουν οι συνάδελφοι, αλλά εγώ αυτό προτείνω. Νομίζω ότι θα ήταν θετικό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Ρομπέρο. καλή ιδέα. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε την πρότασή σου σήμερα το απόγευμα. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Τζιασφέ, η οποία τόσο ευγενικά από το πρωί περιμένει. Θα πρέπει να συζητήσουμε την κατάσταση στο Λίβανο σήμερα το πρωί, αλλά δεν γίνεται πια. Το καταλάβατε, φαντάζομαι κι εσείς. Δεν ξέρω, μπορείτε το απόγευμα να πάρετε το λόγο στις 3, μόλις ξαναρχίσουμε. Α, ωραία γιατί πολύ θέλουμε να σας ακούσουμε, να μας ενημερώσετε όσον αφορά τις διαπραγματεύσει για το σχηματισμό κυβέρνησης στο Λίβανο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που θα είσαστε εδώ. Οπότε ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας για σήμερα το πρωί, το απόγευμα θα τα ξαναπούμε. Το απόγευμα. Ό,τι άλλο θέλετε, το απόγευμα. Να πάμε στο σαλόνι αριθμός 4 του εστιατορίου των ε, μελών στο Ισόγειο. Ε, δεν μου δώσατε το λόγο. Ζήτησα το λόγο από σήμερα το πρωί. Δεν μου έχετε δώσει το λόγο. Πολλά μέλη αντιπροσωπιών δεν μπόρεσαν να πάρουν το λόγο. Ξέρετε, η συζήτηση να έχει πάει μία η ώρα. Όταν ξαναρχίσουμε θα σας δώσω το λόγο. Στις τρεις. Ε, θα είναι αργά.